Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω στη συνάντησή μας. Η συνάντησή μας μεταδίδεται στο ίντερνετ, στο λεγόμενο web streaming. Έτσι θα μπορεί ο κόσμος να δει πώς ε, δίνουμε τη μάχη για τα ανθρωπίνα δικαιώματα järjestyksen. Πριν αρχίσω, παρακαλώ πέστε μου αν εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Esittää lyhyesti tällaisen aikataulusuunnitelman, jota parhaani mukaan koitan noudattaa. Tässä alussa muutamia ilmoituksia lyhyesti. Για να δούμε με δύο λόγια τι θα συζητήσουμε σήμερα, για να σας πω μόνο στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Στη δε συνέχεια, επί μία ώρα, πρόκειται να δούμε πώς έχει κατάσταση στην ε, Βυρμανία. Κατόπιν θα συζητήσουμε για το Αφγανιστάν. Τα δύο τελευταία 45 λεπτά. Θα δούμε τι γίνεται με τις καθηγητήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των βασανιστήριων. Ανακοινώσει του Πρόεδρου πρώτα. Έχουμε την ευρεία ομάδα εργασία, η οποία συναντήθηκε την ε, περασμένη εβδομάδα για να συζητηθεί το πρόγραμμα εργασία για την τρέχουσα θητεία. Είναι κάτι στο οποίο ε, αποτυπώνεται σε ένα έγγραφο το οποίο έχει διαβαστεί σε όλου. Επίση, πρόκειται να ε, γίνει νέα συνάντηση την 1η Οκτωβρίου. Τότε πρόκειται να ληφθεί μια απόφαση για την επόμενη έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Ε, ζητήσαμε τους τονιστές να κατεβάσουν και να προτείνουν ιδέες σε σχέση με αυτήν την ε, έκθεση που θα πρέπει κάποια στιγμή να υποβληθεί εις τους, ε, στη γραμματεία, στο Προεδρείο. Οπότε οι συντονιστέ, όπως ζητήσαμε, πρόκειται να μαζέψουν από τους συνάδελφους ό,τι ιδέε υπάρχουν και έτσι θα δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Στη συνέχεια, να σας πω δύο λόγια για τις ε, αντιπροσωπείες μας, τις αποστολές. Από ό,τι μας έχουν πει, μπορούμε να έχουμε όριο maximum 7 βουλευτών οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις αποστολές αυτές, όσον αφορά τουλάχιστον τη δική μας επιτροπή. Να δούμε τι αποστολές θέλουμε να κάνουμε, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε εκείνες που θέλει έτσι και αλλιώς να προωθήσει το Κοινοβούλιο. και στι αποστολέ αυτέ μπορούμε να στείλουμε δύο δικού μα βουλευτέ. Είναι δε σημαντικό οι συνάδελφοι που συμμετέχουν σε κάποιες ε, αντιπροσωπείες να ενημερώσουν την γραμματεία σχετικά με την γνωστική του συμμετοχή στις αντιπροσωπείες αυτές και όταν ε, πραγματοποιήθηκε αυτή η αποστολή να συμμετέχουν εκεί ως μέλη της Υποπιτροπής μας. Θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα, εάν ήταν δυνατόν, να μπορέσουν αυτοί οι συνάδελφοι να είναι σύνδεσμοι το ΣΥΠΗΝ με τις άλλες αντιπροσωπείες που το Κοινοβούλιο θα πραγματοποιήσει προς διάφορες χώρες. Ακόμα πάντως δεν ξέρουμε τις μερομηνίες. Και όταν μάθουμε τι λεπτομέρειε, τότε μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση για το τι θα γίνει τον Οκτώβριο. έστειλε θέση των Πρόεδρων μια επιστολή σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε σχέση με κάποια κατεπήγοντα του Στρασβούργου για τη, τα απογεύματα την Πέμπτη. Ελπίζω τότε περισσότεροι να προσέρχονται. Εάν ε, δεν συζητούνται πια αυτά τα θέματα τότε και συζητούνται κάποια άλλη ώρα, ποτέ τότε μπορεί να γίνει μια πιο αξιόλογη συζήτηση. Ξέρω, δεν θα είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτή η αλλαγή. Επίσης, ξέρουμε ότι είναι πρόβλημα αυτό, αλλά θα ήταν καλή ιδέα. Όλες οι συνάδελφοι της Επιτροπής αυτό να το ε, γνωστοποιήσουν οι πολιτικές ομάδες ε, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντική υπόθεση για το κοινοβουλίο μας. Άρα θα ήταν καλύτερα να ήταν δυνατόν να γίνει αυτή η συζήτηση. Όχι την πέμπτη απόγευμα, αλλά μια άλλη ώρα. Άρα θα το θέσουμε αυτό στην ε, συνάντηση των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων την επόμενη εβδομάδα. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά την εργασία του Κοινοβουλίου. Όμως, όμως, θα δούμε και κάτι άλλα θέματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τον Μάρτιο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε κείμενο για το Αφγανιστάν, για τις θανατικές ποινές κάποιος για σε θάνατο επειδή έγραψε ένα άρθρο ε, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ισλάμ. Οπότε τώρα κινδυνεύει η ζωή του και άρα θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με κάποιες δολοφονίες ε, ατόμων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα στην Ρωσία. Ο κύριος Μπούζεκ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, απευθύνθηκε στον Υπουργό Εξωτερικών της Προεδρίας της Σουηδίας, τον Καρλ Μπίλτ. Και του ζήτησε να ξεκινήσει κάποιες επαφές και να ξεκαθαρίσει τις ε, απόψεις μας όσον αφορά αυτούς τους ακτιβιστές που τηλεφωνούνται στη Ρωσία. Και το Συμβούλιο όμως αποφάνθηκε σχετικός. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί. Και ελπίζουμε ότι το φθινόπωρο θα γίνουν επαφές περαιτέρω με την Ρωσία. Και αυτό το μήνα θα τα πούμε με τους Ρώσους από αυτό. Και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. Πάντως έχουν γίνει κάποιες ελαφρές αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές ε, έχουν γίνει αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει και θα υπάρξει κάποια ενημέρωση από νομικούς που δικαιούνται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί συζητήθηκε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, στο Στρασβούργο η υπόθεση αυτή. και θα μας πούν όσοι παρέστησαν εκεί τι έγινε. Αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συζήτηση. Αν δεν υπάρχει πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το παριθμόν 3 και αφορά την κατάσταση στην Μιανμάρ. Έχουμε προσκαλέσει στην συνεδρίασή μας τον Χάρν Γιάνγκβε που είναι εκτελεστικό διευθύντη του Euro Burma Office για να μας εξηγήσει για το τι εξελίξει έχουν σημειωθεί και θα δούμε πώς συνεχίζεται η φυλάκιση της Aung San Suu Kyi. Της ε, κυρίας που βραβεύτηκε με το βραβείο Ζαχάροφ. το 1990 της ε, απενεμήθη αλλά έχουμε και πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολείται με τι εξωτερικέ υποθέσει μαζί μα και ένα εκπρόσωπο του ΟΗΕ. Αλλά πρώτος θα λάβει το λόγο ο κύριος ε, Γιάνγκουε για ένα δεκάλεπτο. Και ελπίζουμε να ακολουθήσει κάποια δυναμική συζήτηση με τους βουλευτές και συναδέλφους της Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την Επιτροπή σας, την Υποεπιτροπή σας που μου επέτρεψαν να έρθω. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στην ε, δίκη και τη συνεχιζόμενη κατοίκον κράτηση της Ανσουτσί ε, που δεν μπορεί να αιτιολογηθεί κατά ονδήποτε τρόπο. Η Ανσουτσί έχει περάσει τα 14 από τα τελευταία 20 χρόνια σε κατοίκον περιορισμό και θα έπρεπε στις 27 Μαΐου να λήξει αυτός ο περιορισμός. Ε, μετά από τη λήξη, από το πέρασμα της προθεσμίας δεν υπήρχε άλλος νόμιμος τρόπος για το καθεστώς να την ε, κρατήσει σε κατοίκον περιορισμό. Μετά όμως ένας Αμερικανός ε, πολίτης για το στο όνομα πέρασε στο σπίτι της κυρίας Ανσουτσί κολυμπώντας διέσχισε μια λίμνη για να περάσει εκεί ε, έμεινε δύο νύχτες ε, του επιτράπη να διανυκτερεύσει γιατί ήταν εξατλημένος όπως ισχυρίστηκε και όταν αυτός επέστρεψε κολυμπώντας και πάλι από την άλλη μεριά της λίμνης συνελήφθη και αμέσως μετά η κυρία ε, κατηγορήθηκε ότι παραβίασε τον, το άρθρο 22 του νόμου του 1974, ο οποίος είναι γνωστός ως ο νόμος ο οποίος ε, στόχο έχει να φυλάσει το καθεστώς από ανατρεπτικά στοιχεία. Ο δε νόμος αυτός απαγορεύει την υποδοχή σε κατοίκων περιορισμένους, από κατοίκων περιορισμένους προσκεκλημένων και επίσης δεν επιτρέπει σε άλλο δαπούς να διαμένουν στο σπίτι κατοίκων περιορισμένων. Στις 22 Μαΐου λοιπόν έγινε η δίκη εις βάρος κ. Σανσουτσί. Το δε δικαστήριο επέτρεψε στο, ε, στην κατηγορούσα αρχή να παρουσιάσει 14 μάρτυρες κατηγορίας και μόνο δύο μάρτυρες υπεράσπισης στους ε, συνηγόρους κ. Σανσουτσί. Και λίγο αργότερα καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Η κυρία Ανσουτσί, φυλάκιση η οποία αμέσως μετετράπη από τον πρόεδρο του ε, Κρατικού Συμβουλίου Ειρήνης και Ανάπτυξης σε 18 ε, μήνες κατοίκων περιορισμού με τη δυνατότητα περαιτέρω περιορισμού της διάρκειας αυτής για καλή συμπεριφορά, για λόγους καλής συμπεριφοράς. Με ε, αιτιολογία κατά τη λήψη αυτής της απόφασης ότι η κυρία Σουτσί είναι η κόρη του Αμσάν, του στρατηγού της ανεξαρτησίας και ότι έκανε αυτή τη χειρονομία για το καλό του έθνους. Επίσης μέσα στην απόφαση αυτή υπήρχαν φράσεις ε, όπως ε, προστασία της ειρήνης, της ε, τάξης και της δημόσιας ασφάλειας, να μην υπάρξει ανατροπή της καθεστικής τάξης ή του δρόμου προς τη δημοκρατία κτλ. Η κυρία Σουτσί εφεσέβαλε την απόφαση και η σχετική δίκη στο εφετείο πλέον θα ε, εκδικαστής στις 25 Σεπτεμβρίου, στο Σεπτεμβρίου. Ο Τζον Γετό, εκείνος ο οποίος προκάλεσε αυτή τη νέα ταλαιπωρία για την κυρία Σουτσί, επίσης ε, δικάστηκε, αποφυλακίστηκε όμως επειδή είναι Αμερικανός επίπικος ε, χάρη στη βοήθεια ενός γερουσιαστή ο οποίος μετέβη στη Βυρμανία για να τον βοηθήσει. Η Ανσούκη ήδη βρισκόταν σε καθεστώς κράτησης, ήταν ήδη φυλακισμένη όταν ε, ε, έγινε το επεισόδιο αυτό της παραμονής του Δαπού στο σπίτι της, αλλά δεν είναι δυνατόν να κατηγορηθεί για παραβίαση των όρων ασφαλεία ή κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, διότι η ίδια ήταν κρατούμενη και σχεδόν του δεν μπορούσε να φέρει οδήποτε αντίσταση στο να μπει ή όχι ένα ξένο στο σπίτι τη. Βέβαια, αυτό το οποίο προκύπτει ε, πρακτικά είναι ότι η νέα δίκη θα λάβει χώρα μετά τι προσεχεί εκλογέ και ο θα μπορέσει η κυρία Σουτσίνη να λάβει μέρο στι εκλογέ. Επίση, η βερμανική κυβέρνηση δίνει κάποια σημάδια προς την, ε, προς την κυβέρνηση Ομπάμα επαφές οι οποίες επιτρέπουν στο βιρμανικό καθεστώς να παραγνωρίζει τις επιθυμίες της Κίνας και να ενισχύει τις πιέσεις συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων και καταστολής εις βάρος εθνοτικών μειονοτήτων στα σύνορα με την ε, Κίνα. Πολυάριθμων εθνοτικών ομάδων. Εξαρτώνται βέβαια από την ε, Κίνα, αλλά ε, δεν ήταν ε, το καθεστώς ικανοποιημένο από την εξάρτηση αυτή, γιατί ήταν όλο μεγαλύτερη η εξάρτηση και όλο μεγαλύτερες και οι κινέζικες πιέσεις. Έψαξαν λοιπόν εναλλακτική ως προς την Κίνα και ενώ έκαναν κάποιες προσπάθειες για επαφές στενότερες με τη Ρωσία, τώρα στράφηκαν προς τους Αμερικανούς και αγνοούν τις επιθυμίες των Κινέζων οι δε Κινέζοι δεν επιθυμούν ε, ε, ε, εμπλοκές ή ένοπλες σειράξεις στα σύνορά τους, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν σημαντικές ροές προσφύγων προς την Κίνα σε τέτοια περίπτωση. Ξέρουμε λοιπόν ότι το καθεστώς πιέζει τις εθνοτικές μειονότητες, για τις οποίες ίσχυε καθεστώς κατάπαυσης πυρός τα τελευταία 20 χρόνια, τις πιέζει ε, να υποστηρίξουν στις εκλογές το καθεστώς. Και εάν δεν επιτύχει αυτός ο στόχος, ξέρουμε ότι θα είναι βαριά η καταστολή και βέβαια τα ρεύματα των προσφύγων. Στη δε συνέχεια, η οποιαδήποτε προσπάθεια για αποκλεισμό, εάν συμμετάσχουν οι εθνοτικές αυτές ομάδες στην ε, εκλογική διαδικασία οι οργανώσεις για τη δημοκρατία στη Βερμανία θα μπορέσουν να ισχυριστούν ότι μποϊκοτάρουν τις εκλογές διότι θα έχουν συμμετάσχει όλες αυτές οι ομάδες ε, μειονότητες. Και από την άλλη, εάν μπορέσει αν Σουτσί να είναι ελεύθερη και να συμμετάσχει στις εκλογές, είναι σαφές ότι δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει την εκλογή των δικών του υποψηφίων το καθεστώς. Ε, φυσικά κανείς δεν είναι ικανοποιημένο με, με το στρατιωτικό αυτό καθεστώς στη Βυρμανία και εάν ε, μπορούσε ο λαός να ψηφίσει αυτό που θέλει, να βέβαια ότι δεν θα ψήφιζε το δικατορικό καθεστώς, αλλά υπέρ της δημοκρατίας. Ξέρουμε βεβαίως ότι ο στρατός ε, θα ε, νοφεύσει τις εκλογές του 2010, α, είναι όμως παρόλα αυτά πάρα πολύ σημαντικό να μεριμνήσουμε εμείς να γίνουν στο δυνατόν πιο ε, δικές και ανώθευτες εκλογές στη Βυρμανία, γιατί διαφορετικά χάνουμε για άλλη μια φορά την ευκαιρία να επιτρέψουμε στους ε, πολίτες της Βυρμανίας ε, να εκφράσουν, τη δυνατότητα να εκφράσουν την βούλησή τους. Ο Ταν Σουέ, επικεφαλής του Συμβουλίου Σταθερότητας και Ειρήνης, στρατηγός, στον τίτλο. Έκανε λοιπόν αυτή την ε, περίεργη δήλωση που σας ανέφερα νωρίτερα επειδή η κυρία Ανσουτσί είναι κόρη του στρατηγού Αντσουάν ε, της μετέτρεψε την ε, ποινή σε μονοκατοικό περιορισμό. Με την ομολογία λοιπόν αυτή ίσως αναγνωρίζει ή ίσως υποδεικνύει ότι περιμένει κάποια διαφορετική στάση από την κυρία Ανσουτσί. Δηλαδή, με δεδομένο ότι ο πατέρα τη ίδια θυσιάστηκε αγωνιζόμενο για την ανεξαρτησία του έθνου, ίσω περιμένει και από εκείνη να θυσιαστεί και να αφήσει τι εκλογέ να γίνουν χωρί να παρέμβει, χωρί να ταράξει πολύ τα νερά. σω αυτό σημαίνει ένα νέο καθεστώ, ε, μια νέα τροπή στη Βερμανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μα εξηγήσατε ποια ήταν η κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ανσουτσί και τις συνέπειες που η κατάσταση θα έχει βέβαια στην εκλογική διαδικασία. Ούτως ή άλλως πιστεύω ότι το στρατιωτικό καθεστώς έχει στα χέρια του την εξουσία και δεν είναι εύκολο ε, να παραιτηθεί. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα τον εκπρόσωπο της ε, Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι σε αυτή την συνεδρίαση και μάλιστα πριν από τη συνεδρίαση της Ομάδας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις 6 και 7, ε, στις 26 μάλλον και 27 Σεπτεμβρίου. Εμείς την τον, περασμένο μήνα στην Πανκόκο διοργανώσαμε τη μεγαλύτερη διάσκεψη ε, για την ε, Βερμανία. Ο τίτλος ε, της συνεδρίασης ήταν «Τέλος της ατιμορρησίας στη Βερμανία» και εκεί συγκεντρώθηκαν ε, πολλοί σπουδαίοι εμπειρογνώμονες σε μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια για συζήτηση μελλοντικών στατικικών πριν από τις προγραμματισμένες εκλογές για το 2010. Τα βασικά συμπεράσματα εκείνης της συνεδρίασης ήταν ότι στο διεθνές επίπεδο και στη διεθνή συζήτηση σε σχέση με την πολιτική συμφωλήση, τις πολιτικές εξελίξεις, την εθνική συμφιλίωση και τον εκδημοκρατισμό στην Βυρμανία, το θέμα της ατιμορρησίας και της ε, ε, ε, εγκληματικής λογοδοσίας έλειπε έλειπε και εξακολουθεί να λείπει και σήμερα. Και γι' αυτό και μαζί με τους διάφορους εταίρους μας στην Βερμανία, όπως το Δικηγορικό Σύλλογο της Βερμανίας και άλλους ε, εταίρους, εμείς εκδώσαμε ένα σημείωμα ενημερωτικό σε διεθνές επίπεδο την ημέρα του επανεγκλισμού της Ανσουκή για τα διεθνή εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στην Βυρμανία και την έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής. Ο λόγος της διοργάνωσης αυτής, της, μάλλον της εκπόνησης αυτής της έκθεσης είναι ότι ε, λάβαμε, έχουμε λάβει αρκετές πληροφορίες σήμερα για εκατοντάδες σοβαρών εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, πολεμικών ε, εγκλημάτων, πολέμου μάλλον, ε, και εξακολουθεί η διεθνής κοινότητα να εστιάζει την προσοχή σε πολιτικές εξελίξεις και φυσικά στην ε, κάτοχο του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Και εμείς υποστηρίζουμε τη δουλειά της βέβαια και αποτελεί ένα σύμβολο για τη δημοκρατία στην Βυρμανία. Όμως αυτή η επιλογή για τη δημοσίευση της έκθεσης την ημέρα της ανακοίνωσης της δεν ήταν τυχαία. Λυπούμεθα φυσικά, εκφράζουμε τη λύπη μας για την ατιμιγορία αυτή, ωστόσο θεωρούμε ότι έχουν διαπραχθεί εγκλήματα όχι μόνο στο ανατολικό τμήμα της χώρας κατά των εθνικών μειονοτήτων αλλά και στο υπόλοιπο της χώρας εξακολουθούν ωστόσο οι θύνοντες να μένουν ατιμόρυτοι, να παραμένουν οργανωμένοι ε, μάλλον να γίνονται αυτή τη στιγμή και να διοργανώνονται παρόμοια εγκλήματα από την ε, Χούντα. Θα πρέπει η διεθνής προσοχή να δοθεί με πιο συγκεκριμένο τρόπο σε αυτά τα θέματα και γι' αυτό ακριβώς η FDA ε, το τμήμα της που ασχολείται με τη Βερμανία, συμπεριέλαβε σε αυτή την έκθεση με βάση στοιχεία των Διεθνών Οργανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, για τους εφιάλτες που ζουν καθημερινά οι άνθρωποι της Βερμανίας. Ε, είναι ένα από τα πιο βία καθεστώτα του κόσμου και ο κόσμος βρίσκεται σε δυναμία να επιβάλλει σε μια ομάδα στρατηγών τα διεθνώς αναγνωρισμένα ε, στάνταρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς συνεργαζόμαστε με διάφορους ε, φορείς της ε, Βερμανία αλλά και διεθνείς φορείς. Μεγάλη πλειοψηφία αυτών ε, παρακαλεί και παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστήσει πρώτη προτεραιότητα για την εξωτερική της πολιτική την σύσταση αυτής της Ερευνητικής Επιτροπής πριν από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να επιστήσει τη διεθνή προσοχή στα εγκλήματα που διαπράττονται στη Γερμανία. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των δύο κρατών μελών της που εδράζονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα έπρεπε να ασχοληθεί με πιο δραστήρια και πιο πιεστικά με την άσκηση πίεσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας παρά το σημερινό πολιτικό πλαίσιο το οποίο όλοι γνωρίζουμε. Ε, όλοι είδαμε τα αποτελέσματα της εντυπωσιακής συγκινητοποίησης της ευρωπαϊκής διπλωματίας πριν από την υιοθέτηση του ψηφίσματος για την ε, θανατική ποινή με το μορατόριο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και περιμένουμε ε, τίποτα λιγότερο σε σχέση με τη Βερμανία για, από πλευρά των Ευρωπαίων διπλωματών. Εμείς και διάφορες ε, ενώσεις ε, σύνδεσμοι της Βερμανίας εκφράζουμε τη μεγάλη μας ε, απογοήτευση σε σχέση με τις πρόσφατες κυρώσεις που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από την ετοιμιγορία για την Ανσουκή. Η κοινωνία των πολιτών καθώς και τα δημοκρατικά κινήματα της Βερμανίας ανέμεναν πολύ ισχυρότερη αντίδραση. Αρκετές φορές οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες δικαιολογώντας τη στάση τους ε, για να ξεκινήσουν κάποιο είδος ε, διαλόγου με το καθεστώς λένε πως οι κυρώσεις προφανώς δεν λειτουργήσαν, δεν ήταν αποτελεσματικές, δεν επέφεραν τα αποτελέσματα που, ε, ήταν επιθυμητά. Για την FDA και για τους βιρμανικούς φορείς οι, οι κυρώσεις δεν είχαν καμία επίπτωση γιατί ήταν τελείως ακατάλληλες, είναι ατελείς και άσχημα προσανατολισμένες. Κυρίες και κύριοι, πριν να σταματήσω, θα ήθελα να σας διαβιβάσω ένα μήνυμα από την κοινωνία των πολιτών της Βυρμανίας ε, και από τα δημοκρατικά κινήματα της Βιρμανίας, από τους ανθρώπους δηλαδή που ζουν εντός και εκτός της χώρας και που ελπίζουν για το καλύτερο. Δεν θα πρέπει να πέστε στην παγίδα των εκλογών του 2010. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο θα πρέπει, δεν θα πρέπει να ενθαρρύνει αυτή τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να επιμείνει για την απουσία οποιασδήποτε αξιοπιστία και νομιμότητα της εκλογικής διαδικασία και της αποκαλούμενης ε, ε, δίθεν δημοκρατίας. Η επικύρωση των επικίνδυνου και κακό συντεταγμένου συντάγματος, ε, εκλογέ που έχουν οργανωθεί και που θα γίνουν από το ίδιο το καθεστώ με στόχο να διατηρήσουν την εξουσία τους, και να εγγυηθούν τη θεσμική τους ατιμορρησία σε αυτούς τους στρατηγούς και τα μέλη του στρατού, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι εκλογές δεν αποτελούν καμία, δεν, δεν προσωπεύουν καμία ελπίδα για τη χώρα. Αντιθέτως, όλοι παρατηρούμε και είμαστε μάρτυρες στην κηδεία θα λέγαμε της γερμανικής Δημοκρατίας. Το μάθημα αυτό θα πρέπει επίσης να διαβιβαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους άλλους διεθνείς οργανισμούς, ε, στον ΟΗΕ, στη ΟΣΕΑΝ και σε όλους. Ε, αυτή θα έπρεπε κανονικά να είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τις εκλογές, ενώ είναι υποκράτηση ανσοκή και σταθερά αυξάνονται οι πολιτικοί κρατούμενοι. Υπάρχουν ε, πάνω από 2.200 πολιτικοί κρατούμενοι, ενώ και αρκετά χρόνια η διεθνής κοινότητα καλεί για την απελευθέρωσή τους. Και επιπλέον δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης, ελευθερία του ε, συνέρχεστε, ε, οποιοδήποτε δικαίωμα. Ποιος πραγματικά μπορεί να πιστεύει ότι αυτές οι εκλογές θα είναι δίκαιες, ελεύθερες, καλά διοργανωμένες και ότι ο κόσμος έχει το δικαίωμα να συνομιλήσει και να ε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής διαδικασίας. Ο κόσμος δεν είχε κάνει την ευκαιρία να διαβάσει το Σύνταγμα για το οποίο έπρεπε υποτίθεται να ψηφίσει και μόλις εχθές από τη, στη Χάγη, ενώ εγώ ίδιος ε, ε, συνόδευα υποστηριχτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για της Βερμανία μου έλεγαν ιστορίες ολόκληρων χωριών που καταψήφισαν το Σύνταγμα και το τελικό αποτέλεσμα ήταν υπέρ του Συντάγματος. Με, όχι, με ούτε, ούτε μόνο μία ψήφος κατά δεν ε, υπήρξε για το Σύνταγμα. Την περασμένη εβδομάδα κόσμος ε, συνελήφθη στην Βυρμανία για μόνο και μόνο επειδή είχαν κάποια φέγη βολάν υπέρ της ε, Ιάν Σουκή. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάλογο και η διεθνή κοινότητα απλώ θα, θα, θα μείνει παρατηρήτρια σε μια φάρσα. Σοβαρά εγκλήματα που διαπράττονται εδώ και 40 χρόνια. Πραγματικά συγχωρήστε με για την έντονη γλώσσα που χρησιμοποιώ, αλλά είναι ντροπή για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γιατί αυτό δεν αποτελεί ακόμα ε, πρώτη προτεραιότητα υποστηρίζεται μια ομάδα ανθρώπων που δεν είναι επικεφαλής του κράτους, δεν είναι τμήμα του διαλόγου, αλλά είναι τμήμα του προβλήματος. Αυτή η ομάδα των στρατηγών είναι μια ομάδα εγκληματιών και σε διεθνές επίπεδο έτσι θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, ναι, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλες τις ε, διεθνείς οργανώσεις για τις προσπάθειες που καταβάλουν για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στη Βυρμανία. Ιδιαίτερα απευθύνω λοιπόν ευχαριστήσεις σε εσάς τις ε, οργανώσεις των πολιτών που δραστηριοποιούνται, τις οργανώσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται για να βελτιώσουν την κατάσταση. Ας ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο ή την εκπρόσωπο της Επιτροπής. Αν έχετε την καλοσύνη να μας πείτε τι εξελίξεις υπάρχουν. Μήπως το Συμβούλιο σκοπεύει να επιβάλλει κυρώσεις. Υπάρχει ενημέρωση του Συμβουλίου για αυτή την εκλογική διαδικασία. Θα θέλαμε να δούμε τι απόψη έχει το Συμβούλιο, γιατί δεν πρέπει ασφαλώς να επιβεβαιώνεται η συμπεριφορά της τη χούντας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να σας πω δύο λόγια, να σας αναδείξω τις απόψεις μας, αλλά ιδιαίτερος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, τον Γιάνγκβε. Ε, είναι η φωνή της λογικής, η φωνή της γνώσης και ε, ε, είναι, είναι η ανοχή, η ανεκτικότητα. Είναι κάτι το οποίο όσον αφορά τους εξορισμένους βοηθάει για την συμφιλίωση. Προσέξτε, είναι κάτι το πάρα πολύ περίπλοκο. Εύκολο να πει κανείς, πάμε προς περισσότερες κυρώσεις. ακούμε τα της δίκης, ακούσατε τις ε, απόψεις της Κομισιόν Διαστόματος Μπαρόσο μετά την δίκη, αλλά πρόκειται τώρα και για κάτι άλλο κακό το οποίο έγινε. Είχαμε στην Κόκκαν, στο ανατολικά της χώρας, ε, είχαμε εκεί κάποιες ταραχές και υπήρξε ο κίνδυνος αυτές να επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Επίσης, η υπόθεση αυτή παρέβλεψε και τη σχέση μας με την Κίνα σε σχέση με την κυβέρνηση της χώρας. Και μέσω του ΟΗΕ η Χίλαρη Κλίντον επίσης ανακοινώσε ότι θα αναθεωρήσει την πολιτική της ε, κατόπιν των διπλωματών. Επίσης υπήρξαν και οι ε, προσπάθειες που συνεχίζονται του Γενικού Γραμματεία του ΟΗΕ. Βλέπετε πόσο περίπλοκη έχει καταστεί η κατάσταση και τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα λόγω των κοινωνικών και οικονομικών ε, δυσκολιών. Άρα μια μονοδιάστατη λύση και απάντηση δεν μπορεί να δοθεί. Τώρα, με μηχανικό κατά κάποιο τρόπο η τάση είναι να σωρεύονται οι κυρώσεις. Και αντίστοιχα να διαμορφώνουν και στάση της κυβέρνησης της χώρας. Επομένω, έχουμε εδώ πέρα τώρα τον μποϊκοτάρισμα των εκλογών. Είπαμε να υπάρξει μια στρατηγική μη βία. Οπότε τώρα βλέπετε ότι ο τη πορεία είναι κάτι το διαπραγμάτευτο. Ε, οι στρατηγοί έχουν τα ενία στα χέρια και είχαμε αυτήν την ε, ήσυχη επανάσταση. Επίσης είχαμε όπως είπαμε και τις ταραχές στην Ανατολική επαρχία της χώρας. Οι εκλογέ φυσικά δεν ήταν ελεύθερε, δεν ήταν δίκαιε. Το θέμα είναι τι περιθώρια υπάρχουν να τις κάνουμε δίκαιε και γνήσει τι εκλογέ, αυθεντικές. Από δική μας πλευράς μπορούμε να πούμε ότι μέσω ανθρωπιστική βοήθειας μπορούμε κάτι να κάνουμε. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Υπάρχει περιθώριο επομένω εκεί να σταθούμε. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε και την Ανατολική Επαρχία και ένθεν και εκεί των συνόρων μπορεί να γίνει αυτό η βοήθεια δηλαδή δεν θέλουμε να προχωρήσουμε με σκέτες κυρώσεις θέλουμε μια ισορροπημένη αντιμετώπιση να λάβουμε υπόψη την πολυπλοκότητα της κατάστασης όπως σας προείπα δεν θέλουμε να κάνουμε το κλασικό, δηλαδή την άρνηση του διαλόγου. Θέλουμε να βοηθήσουμε να αλλάξει η κατάσταση. Όσο περνάει από το χέρι μας. Μπορούμε να βοηθήσουμε επομένω ε, με τρόπους ε, κλασικούς. Έχουμε συνομιλητές και Είπαμε να σχηματιστεί ένα ειδικό ταμείο για πολιτισμό, για καλλιεργητές, μικροκαλλιεργητές, ε, αλληλείς. Ένα το πρόγραμμα το οποίο τις αμέσως επόμενες εβδομάδες ή μήνα πρόκειται να ξεκινήσει. Από μόνο τους οι δεν θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η κατάσταση. Αντιθέτως θα επιφέρουν σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης. Πρέπει να μένουν ανοιχτοί οι διεύλοι επικοινωνία. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και αυτό και κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, προσπαθούμε να προχωρήσουμε Προ την υλοποίηση των στόχων της χιλιετία, να δημιουργήσουμε κάποιες νησίδε καλής διακυβέρνηση στη χώρα. Εδώ θα βάλω μία τελεία και ευχαρίστως να απαντήσω ό,τι τυχόν ερωτήσεις έχετε. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε εμείς. Μετά τη συζήτηση να δούμε πώς θα μπορέσει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα όργανα που έχουμε όσον αφορά την ιστορική μας πολιτική. Πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση με του αδέλφου και πέστε μου τώρα ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, έχω δύο ερωτήσει και ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Για τον κύριο Χαν Γιάνκβι, πρώτη ερώτηση. Ο εκπρόσωπος της FDH ε, μας μίλησε για τις εκλογές λέγοντας ότι συνιστά να αντιταχθούμε στην εξαγωγή των ε, εκλογών και να καταδικάσουμε το ότι δεν πρόκειται να είναι ε, νόμιμες ή ανώθευτες αυτές οι εκλογές. Τι περιμένετε ότι μπορεί να προκύψει από αυτό. Και δεύτερη ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από ό,τι μάθαμε επηρεάζει πολύ την ε, κυβέρνηση τη ε, Βυρμανία η Κίνα και το είδαμε αυτό και με την παροχή ανθρωπιστική βοήθεια κατά την ε, φυσική καταστροφή του κυκλώνα που έπληξε τη Βυρμανία αλλά και σε άλλε ευκαιρίε. Πώ σκοπεύετε να συζητήσετε το θέμα αυτό με την κινέζικη κυβέρνηση και του εκπροσώπου τη εδώ ώστε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το τοπίο όπως μας εξηγήθηκε και έτσι ενημερωθήκαμε για την κατάσταση στη χώρα. Φάνηκε έτσι ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την δημοκρατία, τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα του λαού στη χώρα. Αν δούμε τον σχηματισμό μια, ενός μετόπου διεθνούς ε, που θα καταδικάσει την κυβέρνηση της χώρας ακούστηκαν επίσης διαφορετικές απόψεις όπως ε, ακούσαμε και τα αυτά που πιστεύει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μας ζήτησε να είμαστε ρεαλιστές σαν ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τη βάση των όσων ε, έχει χαράξει σαν πολιτική το Συμβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι να υπάρξει συνεργασία και να προχωρήσουμε προς ανθρωπιστική βοήθεια. Νομίζω ότι ε, αναδείται σε ερωτηματικό το τι μπορούμε να κάνουμε εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώπιον αυτή τη κατάσταση. Γιατί η κατάσταση, μα είπε ο υπόσχος Κομισιόν, ότι είναι περίπλοκη, ότι είναι ρευστή. Και είναι τόσο ρευστή που δεν οδηγεί σε κάτι τίποτα το θετικό ως αποτέλεσμα. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε πώς αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση. Ε, η οποία μάλλον είναι τραγικά στατική. Γιατί ε, εντοπίζουμε αυτά τα θέματα εδώ και δεκαετίες. Για την άμμουσα νοσοκία επίσης επιστώνουμε ότι προβληματίζεται την κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από το τέλος δεκαετίας του 80. Πέρασαν τόσα χρόνια και δυστυχώς διεθνής κοινότητα, οι φορείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, κανείς, κανένας δεν μπόρεσε να βελτιώσει την κατάστασή τη. Και δυστυχώ, όπω είπα τη Κομισιόν, από κάθε κρίση βγαίνουν ενισχυμένοι οι στρατηγοί. Και επίση γι' αυτό υπάρχει ο κίνδυνο και από την παρούσα κρίση να βγουν ενισχυμένοι. Συνήθως λέμε ότι όταν παίζεις χαρτιά και δεν είσαι σίγουρος τι να κάνεις να πας πάσο. Σε αυτή την περίπτωση όμως καλύτερα να παρακολουθούμε με επιμονή και υπομονή την υπόθεση και να καταγγέλουμε. Ξεκάθαρα. Οι εκπρόσωποι της ε, ΕΟΚ στον ΟΗΕ, στα διεθνή φόρα και να προσπαθούμε να συνασπίσουμε πείσουμε όσο γίνεται περισσότερους. Να πείσουμε όσο γίνεται περισσότερους. Προς την κατεύθυνση της απομόνωσης της κυβέρνηση της χώρας. Και βέβαια να συνεχιστεί η επαφή με την κοινωνία των πολιτών της χώρας αλλά και να συνεχιστούν τα ενισχυτικά, τα υποβοηθητικά προγράμματα που υπάρχουν. Επομένω, είναι πάρα πολύ έστω αυτό που είπε ο Πρόεδρος να εξαθαρίσουμε ποια είναι η θέση μας, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κοινοβουλίου πριν τις εκλογές. Είδαμε πώς γίνεται η προπαρασκευή, είδαμε τι γίνεται με την αντιπολίτευση. είδαμε ότι η αντιβολή καταγγέλει εκλογές δεν θέλει να κατέβει, να μποϊκοτάρει. Και επεσήμανε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι δεν είναι ούτε ελεύθερε, ούτε δίκαιες οι εκλογέ. Κατηγορηματικά μα είπε αυτά. Η Κομισιόν επομένω θα πρέπει να συμμετάσχουμε θα πρέπει να είμαστε εκεί σαν παρατηρητέ. ή θα πρέπει να το αρνηθούμε λέγοντας ότι πρόκειται για μια εκλογική φάρσα. Δύσκολο το ερώτημα. Γιατί η απλή συμμετοχή των Ευρωπαίων παρατηρητών στην εκλογική τη διαδικασία κατά κάποιο τρόπο τελικά θα νομιμοποιήσει τις εκλογές αυτές. Και είναι κάτι το οποίο μετράει η παρουσία των διεθνών παρατηρητών. Ευχαριστώ. Κύριε Μπιόλς, ο κύριος Κουκάν. Και ίσως μετά να είναι καλό να ακούσουμε και τους ε, προσκεκλημένους μας για να δώσουν τις απαντήσεις. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη που έφτασα με καθυστερήσει τη συνεδρία. Ίσως ήδη να έχουν καλύψει το ερώτημά μου οι διακεκριμένοι προσκεκλημένοι μας, αλλά ας το διατυπώσω. Όπως υπόθηκε λοιπόν, η κατάσταση στη Μιανμάρ δεν αλλάζει. Είναι η ίδια εδώ και χρόνια. Η Aung San με όσο και να έχει προσπαθήσει να τη βοηθήσει όλος ο κόσμος, ε, ταλαιπωρείται ήδη, ταλαιπωρείται ακόμη και παραμένει ακόμη φυλακισμένη. Καθήκον μας λοιπόν είναι να διερευνήσουμε τον καταλληλότερο τρόπο για να της προσφέρουμε βοήθεια και να αλλάξουμε την κατάσταση στη χώρα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων όλων των διεθνών οργανώσεων, με κυβερνητικών οργανώσεων ή ουδήποτε θα μπορούσε να προσφέρει βοήθεια, είναι πολύτιμο εργαλείο. Γι' αυτό και ερωτώ τους προσκεκλημένους που έχουμε τη χαρά να έχουμε μεταξύ μας σήμερα, είναι οι εξής. Ξέρω ότι ο διακεκριμένο καθηγητής Γκαμπάρη από την Νιγηρία και ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών επεσκέφθη την ε, ε Μιανμάρ, αρκετές φορές. Έχει προσπαθήσει να μεταπίσει το καθεστώς, αλλά με μηδενικά αποτελέσματα. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε να αναφέρσουμε υπό την αιγίδα του τον συντονισμό ή εν πάση να δούμε εάν υπάρχουν ήδη προσπάθειες συντονισμού των δραστηριοτήτων αυτών έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτά αποτελέσματα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε πιστεύω να ακούσουμε και άλλη μία σειρά Παρεμβάσω από τους βουλευτές αργότερα, αλλά ας δούμε πρώτα τις απαντήσεις των προσκεκλημένων μας όσον αφορά την εκλογική διαδικασία πρώτα απ' όλα και την Κίνα. Μπορούμε να ζητήσουμε από την Κίνα να στρατευθεί, να έχει τέλο πάντων πιο σαφή στάση έναντι της Βιρμανίας και οι διεθνείς οργανώσεις τι άλλο μπορούν να κάνουν. Παρακαλώ. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει θέμα ε, για τις ε, καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το στρατό και την ανάγκη να σταματήσει η ατιμορρησία με την οποία ε, δρούν. Το θέμα κλειδί, όπως αναφέρθηκε από διάφορους βουλευτές, είναι πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και πώς θα συντονιστεί η διεθνής κοινότητα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι προσπαθώ εδώ και τα 20 χρόνια να φέρω την προσοχή της ε, διεθνούς κοινότητας στη Βερμανία. Η Επιτροπή Euro Burma ε, δημιουργήθηκε για να, να το, η δράση, αλλά όπως ξέρετε η ε, διεθνής κοινότητα δεν έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να σταματήσει αυτά τα εγκλήματα στη Βερμανία. Για πρώτη φορά φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα για αλλαγή εντός της ίδιας της Βερμανίας. Προσπαθούσαμε εκτός τα τελευταία 20 χρόνια. Τώρα για πρώτη φορά λέει ο στρατός ότι θα γίνει γίνουν Η ηρωνία του θέματος είναι ότι θέλουν να κάνουν εκλογέ γιατί πιστεύουν ότι για να είναι θυνομιμοί ακόμα και αν κάνουν απάτη θα πρέπει να δείξουν ότι ο κόσμος τους εξέλεξε. Οπότε το ηρωνικό στοιχείο είναι ότι το δημοκρατικό κίνημα δεν θέλει αυτές τις εκλογές. <laughs> Το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει κανονικά. Δεύτερο είναι ότι δεν συμφωνώ με το Σύνταγμα των Στρατιωτικών. Δεν θέλω να συνεχίσουν να εξουσιάζουν τη χώρα, αλλά αν γίνουν εκλογές, αντί να διοικούν τη χώρα άμεσα ως στρατός θα το κάνουν έμεσα μέσω ενός εκλεγμένου κοινοβουλίου. Φυσικά θα προσπαθήσουν να ελέγξουν το κοινοβούλιο και να χειραγωγήσουν τις εκλογές αλλά απομακρύνονται από την άμεση στην έμεση εξουσία και έχουν επίσης υιοθετήσει την αρχή ότι η άποψη του λαού είναι σημαντική. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν εμείς αυτή την αρχή και να πιέσουμε περισσότερο για αυτή την αρχή ότι δηλαδή η βούληση του λαού είναι σημαντική. Εφόσον όντως έτσι είναι, ας το κάνουμε πραγματικά πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή, να, να, να γίνει πραγματικότητα, πραγματική βούληση του λαού. Εδώ, όπως είπα, σας είπα, 20 χρόνια προσπαθούμε διεθνώς να αλλάξουμε την κατάσταση και δεν τα καταφέραμε. Πώς θα πρέπει από μόνοι μας να αλλάξουμε την κατάσταση. Και το λέω αυτό για το 1990, όταν εξελέγει το κόμμα της Σουκή, εμείς και πολλοί άλλοι, και εγώ ίδιος, γιατί να συγκληθούν εκλογέ, δεν θα είναι δίκαιε και δεν θα είναι ελεύθερε και θα τι χειραγωγήσει ε, το στρατό. Αλλά η σου και αποφάσισε να προχωρήσει σε εκλογέ και ξεκέρδισαν γιατί τελικά την ημέρα των εκλογών μπόρεσαν να ψηφίσει ο κόσμο όπω ε, νόμιζε. Μήπως συμβεί το ίδιο. είμαι σίγουρος πως ο στρατό δεν πρόκειται να τα αφήσει, θα το χειραγωγήσει, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε μήπως και η θέληση του λαού επηρεάσει την κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αν, Αντωνάκη, μπορείτε να κάνετε εσείς τώρα παρατηρήσεις μετά από τα όσα ακούσατε από τους βουλευτές. Just wondering, when we were talking about the failure of international advocacy here, όταν μιλάμε για την αποτυχία του διεθνούς κινήματος, όταν ακούμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχω την εντύπωση πως η αρχή της δική μου παρέμβασης είναι ακόμα κέρια, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ μία στιγμή όπου η καταπολέμηση της ατιμορρησίας στην Βυρμανία έγινε πρώτη προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο και δεν λειτουργήσε. Αντίθετα, η διεθνής κοινότητα επέμενε σε πολιτικό διάλογο, συνδυάζοντας τις, ε, την καλή βούληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Αυτός ο διάλογος ήταν η προτεραιότητα της σημερινής και φυσικά απέτυχε. Σήμερα έχουμε σωρεύσει πολλές αποτυχίες στη Βερμανία και γι' αυτό η FADH μαζί με την, με την ε, κοινωνία των πολιτών της Βερμανίας δεν είμαστε μια εξωτερική οργάνωση που δουλεύει από μακριά για τη Βερμανία. έχουμε μέλη βερμανικές οργανώσεις των πολιτών και εμείς απλώς αποτελούμε το όχημα για τις δική τους, δικές τους Εκεί, αυτοί είναι που δεν επιθυμούν τις εκλογές για ένα πολύ φυσικό και απλό λόγο γιατί εγώ σας έκανα την καρικατούρα του κατά τη διάρκεια της, ομι... μου γιατί θα αποσημάνουν την κηδεία της δημοκρατίας στη Βερμανία. Δεν είναι μια εξέλιξη το να διατηρήσουν ε, ε, έμεσα την εξουσία. Αυτό σημαίνει ότι τους θα νομιμοποιήσουν την εξουσία τους για 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια ακόμα. Αυτό δεν είναι επιλογή για το λαό της Βερμανίας. Θα πρέπει να επανέλθουμε στις προτεραιότητές μας γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι ποτέ υπέρ των κυρώσεων, ε, ιδιαίτερα όταν είναι κατά και του ίδιου του πληθυσμού. Αν λάβετε κυρώσει, αν προβείτε σε κυρώσει, τουλάχιστον προβείτε σε σωστέ κυρώσει. Ε, στοχεύστε το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, τα οικονομικά συμφέροντα. Όλοι γνωρίζουμε ποιε είναι οι εταιρείε που βρίσκονται στη Βυρμανία. Βρείτε λύσεις με τους ασφαλιστές στο Λονδίνο. Το, κέντρο, το Διεθνές Κέντρο για τις Ασφαλίσεις είναι το Λονδίνο, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάντε συνολικέ κυρώσει και σταματήστε όλου από το να μπουν στη Βερμανία, ακόμα και του Κινέζου ή του Ινδού. Ε, θα πρέπει κάποια στιγμή να τα πούμε έξω από τα δόντια δεν υπήρχε πολιτική βούληση ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπλοκάρει τελείω την πρόσβαση των Βυρμανών στρατηγών στην τράπεζά τους, στις τράπεζές τους. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Και δεύτερον, η περιπλοκότητα της κατάστασης στη Βυρμανία είναι πραγματικά πολύ πολύ ε, ευαίσθητη. Αλλά το ίδιο ισχύει για την Ταρφούρ, την Κολομβία, το Κονγκό. Γι' αυτό οι διεθνεί οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπω η δική μα, η FIDH, στηρίζουν τα τοπικά κινήματα. Είναι δική του η χώρα. Και εκείνοι ξέρουν ποια είναι η κατάσταση και πόσο περίπλοκη είναι, πολύ καλύτερα από ότι άλλοι εκτό. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να μιλάμε για εκλογές. Αφού ο κόσμο τι κάνει και γνωρίζει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι πολύ, πολύ περίπλοκο με διάφορα επίπεδα κοινοβουλίου, σώματα από εδώ, από εκεί, δεν θα αφήσουν τον κόσμο να υπάρξει διάλογο. Επανέρχομαι στο ίδιο. Πώς περιμένετε να γίνει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη σε, μια, ένα από τα πιο βία καθεστώτα του κόσμου. Θα πρέπει να αναζητήσετε άλλη επιλογή, να κάνετε πολιτική διάλογο, αλλά από τη στιγμή που θα έχετε αρχίσει να αντιμετωπίζεται το θέμα της ε, λογοδοσίας των εγκληματιών. Και αυτή θα πρέπει να είναι ο αγώνας κατά της ατιμωρησίας. Δεν έχει ξεκινήσει καν αυτός ο αγώνας. Και μετά μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε κύριε Αθανασίου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 η συνεδρία στο ΑΣΕΜ e θα γίνει εδώ στη Βρυξέλλο στο Σεπτέμβριο του 2010. Πώς που το προβλέπετε εσείς αυτό στη Βερμανία ε, με βάση αυτή την ε, διάσκεψη κορυφής εδώ στις Βρυξέλλες. Και αυτό το ερώτημα απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε ένα φόρουμ ταυτόχρονα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε το Κοινοβούλιο να το δεχτεί. Εγώ ε, σας είπα ότι ότι κάθε εβδομάδα, κάθε φορά συγγνώμη, συμμετέχω στις συνεδριάσεις αυτής, ε, για αυτές τις χώρες. Ο υπουργό Εξωτερικών της Φιλανδίας θυμάμαι ότι είχε αντιμετωπίσει μια χώρα ε, όπως η Βερμανία. Είχε έρθει εδώ και εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης της Βερμανίας. Ίσως μπορούμε να το κάνουμε αυτό την επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Βυρμανία είναι πλήρως μέλος της ασιατικής πλευράς του ΑΣΕΝ, άρα μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις που γίνονται στην Ευρώπη. Όμως, το να είναι παρούσα η κυβέρνηση της Βερμανίας μέσα στην, ε, στο ΕΣΕΝ είναι καλύτερη επιλογή από το να τους απομονώσουμε γιατί η απομόνωση ωφελεί την κυβέρνηση. Αγα, ε, της αρέσει η απομόνωση για να συνεχίζει να κάνει το δικό της ε, χωρίς τον έλεγχο του διεθνούς κοινότητας. Ε, τώρα με την Κίνα. Η πίτροπο μου, η κυρία Φερέρο Βάλτνερ, είναι προσωπικά δεσμευμένη να αναφέρει τη Βυρμανία σε κάθε πιθανή περίπτωση και το κάνει αυτό τακτικά στις συναντήσεις της με τους Κινέζους. Επίση, επίσης αναφέρεται διαρκώς η Βυρμανία στο πλαίσιο της ε, ε, ΑΖΕΑΝ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κάθε φορά που υπάρχει τέτοια συνάντηση και όλες οι εξελίξεις οφείλονται εν μέρη στην επιμονή μας στο θέμα. Έχουμε έναν ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον χρησιμοποιούμε και καθε... διαρκώς η κυρία Βάλτνερ ε, παροτρύνει την κυβέρνηση της Βυρμανίας, της Μιανμάρ να έρχεται σε επαφή με τον κύριο Φασίνο που είναι ο ειδικός απεσταλμένος. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για την Βυρμανία. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ομοιόμορφη στάση. Είναι πολύ καλό που έχουμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις και που πολύ ε, στεναρές γραμμές ακολουθούν. Σαφώς και η κατάσταση δεν είναι σταθερή. Φαίνεται να είναι σταθερή, αλλά υπάρχει μετάβαση. Υπάρχει ένας ε, οδικός χάρτης, η κατάσταση όπως σας είπα είναι ρευστή και περίπλοκη. σε ένα χρόνο θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τον απόφευκτο. Θα υπάρχει μια ατελής αλλά εκλεγμένη κυβέρνηση. Γίνεται, είναι, είναι μια αλλαγή σε εξέλιξη. Οι πιθανότητε ε, να υπάρξει επιτροπή παρατήρηση εκεί από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απίθανε, είναι πολύ λιγοστέ. Ε, και αυτό πρώτον γιατί η κυβέρνηση θέλει να είναι απομονωμένη, έπειτα θα έχουμε το θέμα του να νομιμοποιήσουμε την κατάσταση ή όχι, αλλά το βασικό θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να βλάβουμε πρόσκληση για να υπάρξουν παρατηρητέ. Η κυβέρνηση αορίστως είπε ότι μπορεί να επιτρέψει σε διπλωμάτες του ΑΣΕΑΝ να έρθουν ε, για λίγο χρονικό διάστημα ως παρατηρητές. Τέλος, για την, ε, τις διάφορες φωνές που ακούγονται εντός της ε, χώρας. Από τα πολυορίθμα μου ταξίδια έχω πάει στη χώρα περίπου 38 φορές αν μετρήσω τις θεωρήσεις μου, τις φραγίδες μου στο διαβατήριό μου Δεν άκουσα ποτέ τόσο διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, πολύ διαφορετικές για τις εκλογές. Υπάρχει μια ομάδα που είναι υπέρ της κυβέρνησης και που θέλει να θεσμοποιήσει, να θεσμοθετήσει ένα υβρίδιο σύστημα κυβέρνησης ανάμεσα στο στρατιωτικό και τους πολιτικούς ε, για να μπορέσει να κυβερνήσει. Υπάρχει μια άλλη ομάδα εθνοτική που δεν είναι δημοκρατικά νόμιμη και θέλει να νομιμοποιηθεί μέσω των εκλογών ε, και έπειτα υπάρχει μια τρίτη ομάδα που συνεχίζει ένα είδος ε, στάνταρ γραμμής ε, αντιπαράθεσης ό,τι και αν λέει η κυβέρνηση είναι λάθος, αυτό είναι Αυτή είναι η γραμμή την οποία ανέφερε ο Γιάνγκ δηλαδή η αντιπαράθεση. Και έπειτα υπάρχει και μια τέταρτη ομάδα που υποστηρίζει το να μπουν στην, στον οδικό χάρτη ως αξιόπιστα άτομα που θέλουν να δουλέψουν εντός του συστήματος. Βλέπετε λοιπόν ότι η στάση του κόσμου, ακόμα και μέσα δηλαδή στην ε, Βερμανία, είναι πολύ διαφοροποιημένη και ειλικρινά και θα έλεγα ποιοι είμαστε εμείς να πούμε στην κοινωνία των πολιτών της Βερμανίας τι να σκεφτεί για τον οδικό της χάρτη. Είμαι πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο τόσο ώστε να συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Κύριε Νίλσεν, θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Για πετε μας. Τι γίνεται με αυτά τα πέντε σημεία. το για ένα πρόγραμμα δράση που είχε προτείνει ο κ. Καμπάρη. Πώς γίνεται το θέμα. Επίσης, ένα ερώτημα προς την FDH. Είχατε δει, είπατε ότι θέλετε να συγκροτηθεί μια διεθνής επιτροπή σε σχέση με τα ε, εγκλήματα τη ανθρωπότητα και ξέρουμε ότι δυστυχώ τα τελευταία χρόνια διεθνώς γίνονται τέτοια εγκλήματα. Εσείς επομένως ε, τι προσδοκάτε από αυτήν την επιτροπή που συγκροτηθήκε. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Νίλσεν. Ο κύριος Γιάνγκβε νομίζω πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση που υποβάλλατε. Έχετε το λόγο κύριε Γιάνγκβε niin, nyt ymmärrän, että se oli enemmän osoitettu herra Atanasiolle, mutta muutkin voivat toki kommentoida. Herra Atanasio, olkaa hyvä. ίσως ε, την Αθανασίου. Ίσως εκείνος πρέπει Je vais commencer avec la Commission internationale d'enquête parce que c'est beaucoup plus facile dans les sens où... Να μιλήσουμε για την Διεθνή Ερευνητική Επιτροπή. Γιατί ξέρουμε το περιβάλλον το πολιτικό στο οποίο δουλεύουν ε, οι διπλωμάτες και οι μη κυβερνικές οργανώσεις. Οπότε ας ξεκινήσουμε με αυτή την Διεθνή Ερευνητική Επιτροπή. Αν δείτε την ε, ε, έκθεση, παραπέμπει στα άρθρα 7 και 8 του καταστατικού όπου τα εγκλήματα από εκεί που προβλέπονται γίνονται στην Βυρμανία. Και δεν ζητήθηκε δεν ζητήθηκε παραπομπή στο διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Γιατί αυτό θα τον μπλοκάριζε το Συμβούλιο ασφαλή του ΙΕ. Γι' αυτό και προχωρήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Με τη Διεθνή Ερευνητική Επιτροπή, τόσο ώστε στο Συμβούλιο ασφαλή να περάσει το μήνυμα. Λοιπόν, να πήραν αυτές τις πληροφορίες. Άλλωστε είναι αλήθεια ή μία αλήθεια. Αλλά υπάρχουν εδώ πέρα ενδείξει ότι, ότι τελούνται κλίμακα τη ανθρωπότητα εκεί. Και είπαμε ότι θα πρέπει να ασχοληθεί αυτή η επιτροπή και να δούμε τι ισχύει. Ίσως αυτό κάτι αποδώσει στο Συμβούλιο Ασφαλεία, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι τη ε, υποστήριξουν αυτή την πρωτοβουλία, γιατί θα χρειαστεί επομένω μια δυναμική βοήθεια από ΕΕ, από Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα άλλα μέλη τη Συμβουλίου Ασφαλεία. η δε πολυμορφία, η δε ποικιλία που υπάρχει στην, ε, στην Ασία, γιατί διευθύνει το λογαριασμό του FDH, ε, έχει να κάνει με αυτό που λέμε αξίες της Ασίας. αυτό το καταστατικό της Ρώμης, του, του Διεθνούς Πυρηνικού Δικαστηρίου, το οποίο δέχεται την αρχή του ότι υπάρχουν κάποιε αξίε στην αξία διαφορετικέ και γι' αυτό λέμε ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι η νομική προσέγγιση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με την τιμωρησία, τι θα γίνει με την ε, χώρα σε μια. Με την υγεία ειρήνη σε μια χώρα, γιατί ε, δεν είναι δυνατόν αν έχουμε θεσμοθετημένη αντιμορφή σε μια χώρα να έχουμε ειρήνη. Θα πρέπει όλοι να, να, να το έχουμε αυτό υπόψη, να το θυμόμαστε πάντα. Και καταλήγω κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει να απαντήσω στα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ δεν μιλούμε για κάποια κυβέρνηση. Μιλούμε για κάποια ομάδα στρατιωτικών οι οποίοι ε, κρατούν εχμάλωτη μια χώρα. Βεβαίω και χρειάζεται συνομιλητή όσον αφορά του διπλωμάτε μα, τη δική μα πολιτική, αλλά δεν πρόκειται περί κυβερνήσεων, πρόκειται περί ομάδα στρατηγών. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, το οποίο επίση δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και θα πρέπει να ε, χαράσουμε την πολιτική μας έχοντας πάντα υπόψη κάτι τέτοιο. Και δεν είναι το θέμα το κατά πόσο θα, τους πούμε των Βυρμανών πώς θα ε, δικούν τη χώρα τους. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ σε κάποιο διεθνές φόρουμ. Η FDH συνεργάζεται με τους Βερμανούς. Ακόμα και αν ε, είμαι Έλληνας και εγώ όπως και ο συνομιλητής μου έχω περάσει όλη τη ζωή με τους Βερμανούς και ε, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι υπάρχουν προσδοκίες από το δημοκρατικό κίνημα ε, όσον αφορά το τι θα κάνει η διεθνή κοινότητα. Και το λένε. Χρειάζονται την υποστήριξή στη βοήθειά σας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μην αρνηθούμε την βοήθειά μας επί τη βάση της πολιτικής που εκείνοι μας προτείνουν το δημοκρατικό κίνημα της χώρας που δεν το να λέμε ότι παρότι είμαστε έξω από το χώρο ξέρουμε καλύτερα τι γίνεται με την διεθνή διπλωματία δεν, δεν είναι εδώ θέμα καν άσκηση διπλωματίας είναι θέμα προστασίας των δικαιωμάτων ενός λαού αυτή είναι, αυτή θα έπρεπε να είναι η αφετηρία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον κάθε διεθνή φορέα που θέλει να ασχολείται με την ειρήνη και τη σταθερότητα στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αγγουέ, θα θέλατε παρακαλώ και εσείς ε, να διατυπώσετε τις παρατηρήσεις σας για την ατιμορρησία ή για κάτι άλλο, αν ενδεχομένως έχετε να προσθέσετε. Παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει διαφωνία με τα όσο προσπαθεί να κάνει το FIDH. Το πρόβλημα είναι ότι οι δικές τους προσπάθειες είναι μάλλον μακροπρόθεσμες, χρόνο, ένα μακροπρόθεσμο εγχείρημα. 10-20 χρόνια αργότερα να δούμε τα αποτελέσματα. Οι εκλογές όμως είναι του χρόνου. Και κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν αρκεί να πούμε ότι μποϊκοτάρουμε ότι απέχουμε από τι εκλογές, ε, γιατί είναι υποχρεωμένο ο καθένας να λάβει μέρος σε εκλογές στη Βυρμανία. Είναι υποχρεωτική ψηφοφορία. Και δεν υπάρχει θέμα νόθευση ε, νοθείας στι εκλογές. Γιατί εάν πάει ο κόσμος να ψηφίσει, αναγκαστικά θα ψηφίσει το κόμμα των στρατιωτικών, εφόσον δεν συμμετάσχει η αντιπολίτευση. Και μπορούμε εμεί εδώ πέρα, όταν ερχόμαστε στην Ευρώπη, να λέμε ναι, δεν ήταν οι συνθήκε ισότιμε για τη συμμετοχή τη αντιπολίτευση, αν απόσχει από τι ε, εκλογικέ διαδικασίε η αντιπολίτευση και δεν ήταν σωστέ οι εκλογέ. Αλλά οι Ασιάτε και οι γείτονε τη Βυρμανία, τα γειτονικά κράτη, θα πούνε μα δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκλογέ έγιναν, ελεύθερε ήταν, αποτέλεσμα βγήκε και ψηφίσανε το καθεστώ. Σε αυτό θα πρέπει να αντιδράσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Λέει η Πρόεδρος. Η συζήτηση γιατί η Βυρμανία ήταν πολύτιμη, πολύ χρήσιμη. Θα τη συνεχίσουμε ασφαλώς και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολύ σύντομα μάλιστα, γιατί θα έχουμε την ε, ε, συνεδρίαση με τα κράτη της ΝΑΖΑ και νομίζω ότι θα αποτελέσει αυτή την ε, καλή ευκαιρία να εξετάσουμε τις ε, προοπτικές, τις στρατηγικές που μπορούμε να υιοθετήσουμε. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλους τους προσκεκλημένους μας για τις παρεμβάσεις και την παρουσία σας εδώ. Ξέρω ότι ενδεχομένως έχετε διαφορετική στρατηγική μεν και ιδέ. Παρά τις διαφορές όμως αυτές αγωνιστήκατε κατά τρόπο ειρηνικό μαζί μας. Συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτή την ε, συζήτηση και εμείς με την Κομισιόν αλλά και με το Συμβούλιο. Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Αλλά τώρα ας περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης το Αφγανιστάν. Valiokunnan puheenjohtajan Eva joka istuu eh, huoneessa. θα καλωσορίσω εδώ τους εκπροσώπους που έχουν έρθει να μας μιλήσουν για την κατάσταση του Αφγανιστάν μετά τις εκλογές. Το θέμα ξέρω ότι το είδατε την προηγούμενη εβδομάδα και το σύστησατε και στην Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων. Ασφαλώς η σημερινή συζήτηση δεν θα είναι η τελευταία για το Αφγανιστάν. Ακούσαμε ανησυχητικές αναφορές και εκθέσεις για την κατάσταση των ανθρωπινών δικαιώματων ε, στη χώρα αυτή. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Αχμάτζη Αλάγκαρη μέλος Ανεξάρτητης Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αφγανιστάν. Με μεγάλη χαρά λοιπόν σας βλέπουμε εδώ και εσάς αλλά και την κυρία Ρετσέλου Ρίντινγκ από το Human Rights Watch που ήρθε από την Καμπούλ και αυτή για να μας μιλήσει. Έχουμε εκπρόσωπο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, David Ells το όνομα, που ασχολείται με τα θέματα της πολιτικής έναντι του Αφγανιστάν και ο οποίος, αν δεν απατώμε, έχει πολλά μίλια κάψη μεταξύ Καμπούλ και Βρυξελών. Και ξέρετε ότι υπάρχει αντιπροσωπεία στο Αφγανιστάν υπό τον στρατηγό Μοριγιών βέβαια στο Αφγανιστάν. Παρακαλώ λοιπόν να λάβετε το λόγο. Έχει το λόγο κυρία Αχμετζία Λάγκαρη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζιαλάνγκαρη, παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Εσείς, ο κύριος Λάγκαρη θα μιλήσει πρώτος. Ναι, ναι, παρακαλώ. okay, eh? good morning everyone. Uh, I'm very happy that I'm being here and... Uh, Καλημέρα σας. Ευχαριστώ τους αξιότιμους ευρωβουλευτές για την τιμή που μου κάνουν και την προσοχή που δίδουν στο πρόβλημα που έχουμε στο Αφγανιστάν μου εξασφάλισαν τα έξοδα ταξιδιού για να έρθω να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, πράγμα το οποίο δείχνει πόσο πραγματικά και ειλικρινά ανησυχούν. Η κατάσταση ανθρωπιστική στο Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή είναι ανησυχητική. Είναι πολλά τα προβλήματα προς την ασφάλεια λόγω των απειλών των τρομοκρατών και τα λιμπάνα, αλλά συγκρινόμενοι με το 2002 ασφαλώς ε, παρουσιάζει πολλές εξελίξεις και ως προς την ελευθερία του λόγου και ως προς τα δικαιώματα των γυναικών. Και ως προς ε, την αντιμετώπιση των δικαιωμάτων των ε, ατόμων με αναπηρίες. Πολλά πράγματα εξελίσσονται προς το καλύτερο στο Αφγανιστάν. Δραστηριοποιείται τώρα η κοινωνία των πολιτών οι πολίτες μπορούν να μιλήσουν και να εκφράσουν τις θέσεις τους, ενώ 4-5 χρόνια πριν ακόμα δεν μπορούσαν να το πράξουν αυτό. Πολλά υποσχόμενα λοιπόν αυτές οι εξελίξει, αλλά παραμένει ανησυχητική η κατάσταση ακόμα. Ένα πράγμα το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι κάποιος ο οποίος είχε συλληφθεί πέρυσι για την ε, θέση κυκλοφορία ενός, μάλλον για την διάθεση κάποιων φίλων του ενός κειμένου που είχε κατεβάσει από το ίντερνετ γιατί ήταν υποτίθεται προσβλητικό προς το Ισλάμ. Αυτός ο άνθρωπος φυλακίστηκε για αρκετά χρόνια μάλιστα και καταδικαστεί, αλλά ευτυχώς πριν από λίγο ακόμα, πριν από λίγες μέρες, αποφυλακίστηκε. Έμεινε για λίγες μέρες στην Καμπούλ και από ό,τι μάθαμε από τις εφημερίδες αποχώρησε από τη χώρα εντωμεταξύ, δεν ξέρουμε ακριβώς, που βρίσκεται. Έτσι βλέπουμε ότι οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητες και οι πιέσεις που ασκήθηκαν στην κυβέρνηση για την αποφυλάκηση αυτού του ε, νεαρού και βέβαια οι προσπάθειες και της δικής μας Επιτροπής όπου είχαμε προσωπικές επισκέψεις στη φυλακή στον άνθρωπο αυτόν, αλλά και συλλογή ε, υπογραφών, πάνω από χίλιε υπογραφές υπέρ τη αποφυλαξής του, έφεραν καρπούς από ό,τι φαίνεται. Uh, uh, Ξέρετε ότι έγιναν οι ε, εκλογές ε, για την θέση του Προέδρου αλλά και οι περιφερειακές εκλογές τον Αύγουστο και η κατάσταση παραμένει πολύ ασαφής, αβέβαιη και ανησυχητική. Οι εκλογές λοιπόν με το και μόνο η διεξαγωγή των εκλογών πρέπει να πούμε τον Αύγουστο ήταν με όλα αυτά τα προβλήματα και την ανασφάλεια που επικρατεί ήταν επίτευγμα το ότι ο κόσμος πήγε στις κάλπες, το ότι έλαβε το θάρρος να συμμετάσχει στις εκλογές. και από το 74,2% των ψήφων που καταμετρήθηκαν, 3.908.335 ψηφίσαντες δηλαδή, από ό,τι λέει η Αφορευτική Επιτροπή, το 31% δεν έχω ακριβώς τον αριθμό, ε, ήταν γυναίκες ψηφοφόροι. Πολύ ικανοποιητική λοιπόν εξέλιξη. Είχαμε συνολικά 221 221.446 ε, παρατηρητές από 2.972 ε, οργανώσεις, διεθνείς οργανώσεις, οργανώσεις πολιτών, περιφερειακές που είχαν πάει ως παρατηρητές των εκλογών στο Αφγανιστάν. Όλοι αυτοί οι παρατηρητές λοιπόν από όλους αυτούς 61.951 ήταν οι γυναίκες. Οι λοιποί ήταν άνδρες. Να σας δώσω μερικά στοιχεία για τις εκλογές που εκλήθηκαν σε δύσκολες συνθήκες και δυστυχώς είναι λυπηρά τα νέα. Είχαμε επί παραδείγματι την ημέρα των εκλογών εκρήξεις βομβών σε διάφορα σημεία, σε ένα ε, ε, αστυνομικό τμήμα μπροστά, σε δύο σημεία στην Καμπούλ. Επίθεση από τρομοκράτες στις βάρος αστυνομικού τμήματος στην Καμπούλ. Άλλα πράγματα, αντίστοιχα φαινόμενα έχουμε και στο βορρά του Αφγανιστάν, επιθέσεις εις βάρος εκλογικών τμήματων, επιθέσεις με, πύραυλος, με πυράβλους σε πολλές επαρχίες με των οποίων και Κανταχάρ. 50 περίπου ήταν τα θύματα αυτών των επιθέσεων, εκ των οποίων μισή είναι τα 130 οι επιθέσεις συνολικά ε, με πύραυλο, είτε επιθέσεις αυτοκτονίας, ε, βομβιστικές επιθέσεις, με πολλούς νεκρούς και τραυματίες εκείνη την ημέρα. Εννέα ήταν οι πολίτες και 11 τα μέλη των φορευτικών επιτροπών που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα. Από τις ε, ε, από τις ε, επιθέσεις μεταξύ των οποίων οι έξι ήταν και βομβιστικές, ήταν επιθέσεις αυτοκτονίας, 50 απετράπησαν κατά τη διάρκεια των εκλογών. Το δε Αύγουστο με την προετοιμασία των εκλογών 32 στρατιώτες Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους, 4 οι Βρετανοί, ...21 Ταλιμπάν που σκοτώθηκαν Πολλά είναι τα δεδομένα που έχουμε να παρουσιάσουμε. Παρόλα αυτά όμως, παράλληλα αυτή την έκθερη ρυθμή κατάσταση, οι πολίτες προσήλθαν στις κάλπες. Και θα επαναλάβω, υπήρξαν ε, κακοδιαχειρήσεις των εκλογών, υπήρξαν παραβιάσεις νομοθεσίας, προβλήματα σε διάφορα εκλογικά κέντρα. Ένα εκλογικό κέντρο μάλλον, μάλιστα ούτε καν άνοιξε, οι κάλπες του όμως πήγαν στο άλλο, σε κάποιο άλλο εκλογικό κέντρο γεμάτες με ψήφους. Και σε, κάποιο, σε κάποια από τις κάλπες ε, ανακάλυψαν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ότι είχε μπει ολόκληρο το πακέτο, το μπλοκάκι δηλαδή των ε, ψηφοδελτίων, χωρίς καν να κάνει κανείς τον κόπο να ξεχωρίσει τα φύλλα, όλο το μπλοκάκι όπως ήταν ενωμένα, το είχαν ρίξει μέσα στην κάλπη. Υπέρ ενός εκ των υποψηφίων. Και πρέπει να σημειώσω εδώ ότι δεν ε, είχε ιδιαίτερη μεταχείριση ένα μόνο υποψήφιο. Δηλαδή αυτέ οι παρατυπίε συνοθείε δεν έγιναν μόνο υπέρ ενό υποψηφίου. Έγιναν υπέρ διαφόρων, διαφορετικών ε, στρατοπέδων. Πριν από τις εκλογές επίσης ε, με την προετοιμασία, την επιμελητιακή θα έλεγα προετοιμασία, η οποία ήταν ικανοποιητική. Ε, έγινε λοιπόν η οργάνωση όπως είπα, μεταφέρθηκε το υλικό για τις εκλογές στα εκλογικά κέντρα, σε ορισμένα όμως δεν κατέστη δυνατό αυτό. Ορισμένα δεν άνοιξαν καν για λόγους ασφαλείας. Και επίσης πολλά προβλήματα ε, μπορεί να υπήρξαν, αλλά πρόοδος σημειώνεται. Πριν από τις εκλογές τώρα, για να επανέλθω, έγινε προσεκτική μελέτη της κατάστασης από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ε, λάμβανε και διαμαρτυρίες ως προς τις ε, προεδρικές εκλογές όπως και για τις περιφερειακές εκλογές. και ε, κηρύχθηκαν ως μη ε, εκλόγιμοι, δηλαδή απεκλείστησαν τις εκλογικές διαδικασίες ορισμένοι από τους υποψηφίους περιφερειακές εκλογές. Πρέπει να πω ότι είχαμε μάλιστα δύο γυναίκες ε, υποψήφιες αντιπροέδρου σε περιφέρεια εν προκειμένου δείγμα θετικό για την εξέλιξη της κατάστασης αλλά δυστυχώς δεν εξελέγησαν, δεν είχαν ικανοποιητικό αριθμό ψήφων. Επίσης ανησυχητικό είναι ότι ορισμένοι υποψήφοι δεν είχαν στη θέση τους αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν την προεκλογική τους εκστρατεία Κάποιοι, λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι μπόρεσαν να συλλέξουν επαρκή πόρους για να αναπτύξουν την εκστρατεία τους μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κάποιοι, ο λιγότατοι, δύο ή τρει μπόρεσαν να δαπανίσουν μάλιστα πολλά χρήματα προβαλλόμενοι και στα τηλεοπτικά κανάλια κατά τι ώρες της μεγάλης ε, τηλεθέασης. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ένα λεπτό προβολή στην τηλεόραση κοστίζει 600 δολάρια στο Αφγανιστάν. Την ώρα εχμής. Κάποιοι λοιπόν μπόρεσαν να, δαπανίσουν μέχρι, να εξασφαλίσουν μέχρι και μία ώρα τηλεθέαση ή μισή ώρα προβολή στην τηλεόραση. Επίση, προβλήματα υπήρξαν ω προ τη δυνατότητα για ορισμένε γυναίκε να μεταβούν στι ε, περιοχέ, να πάνε από σπίτι σε σπίτι και να μιλήσουν με του ε, πολίτε προβλήματα είχαμε ε, και στο επίπεδο ορισμένων υποψηφίων ε, που υπέστησαν επιθέσεις, μάλιστα ένας από αυτούς έχασε τη ζωή του. Προβλήματα λοιπόν, επιθέσεις, εκφοβισμός υπήρξε. Είναι όμως για μας τεράστιο επίτευγμα το ότι έλαβε χώρα η εκλογική αναμέτρηση. Και πρέπει βέβαια αυτό να το αναγνωρίσουμε. Τώρα πια πρέπει να δούμε βέβαια, και αυτό είναι το πρόβλημα, το πώς θα χειριστεί η Εφορευτική Επιτροπή το, τις 600 και πάνω διαμαρτυρίες ενστάσεις επί των εκλογών. Άρχισε λοιπόν η καταμέτρηση εν μέρη από την Εφορευτική Επιτροπή. Όμως μετά άρχισαν οι ενστάσεις από τους υποψηφίους που έλεγαν ότι δεν υπάρχει διαδικασία για την αντιμετώπιση των ενστάσεων και είπανε καλύτερα θα πρέπει να γίνει πρώτα επεξεργασία όλων των ενστάσεων, να δοθεί απάντηση σε κάθε ένσταση χωριστά και μετά να γίνει η καταμέτρηση. Η Επιτροπή Εφορευτική αποφάσισε να προχωρήσει σε μερική έστω καταμέτρηση. Μετά τι διέκοψε και εν αναμονή της ε, επεξεργασίας και διερεύνησης όλων των ενστάσεων σταματάει η διαδικασία, διακόπτεται και θα συνεχιστεί όταν έχουν δοθεί απαντήσει σε όλες τις ενστάσεις. Ευχαριστώ. Αυτά είχα να πω προς το παρόν και περιμένω τις παρατηρήσεις ή ερωτήσεις των βουλευτών. Ε, Συνεχίζουμε. Η ενημέρωση θα γίνει τώρα την κυρία Τζορβίτ. Έχετε το λόγο. Δουλεύει τα μικρόφωνα, μάλιστα. Σα ευχαριστώ που με καλέσατε για άλλη μια φορά και για που οργανώσατε αυτή την ακρόαση. Ε, όλα όσα είπε ο προλογητή σα τα πήρα πάρα πολύ αξιόλογα. Σα μιλήσω και εγώ για τι εκλογέ αλλά και για τα δικαιώματα των γυναικών και επίση το πρόβλημα τη ε, ατιμορρησία και όποιο έχει τυχόν ερώτηση μπορεί να την υποβάλει στη συνέχεια. Ακριβώς όπως ε, ελέγχθη, πρόκειτο για πάρα πολύ βίαιη περίοδο γιατί είχαμε πάρα πολλά επεισόδια σε όλη τη χώρα. Τελευταία τα τελευταια είναι 7-8 τις πιο α, βίαιες ε, εκλογές και ημέρες. Α, αυτό φυσικά είχε σημασία σε νότρα τελικά τη χώρα ε, όσον αφορά την συμμετοχή σε εκλογέ. Είχαν πάρα πολύ μεγάλη εποχή κυρίω των γυναικών λόγω τη βία και αυτό επίση έστω στον δρόμο για νοθεία μεγάλη, ιδίω ε, στι περιοχέ που υπάρχουν συγκρούσει. Δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ εκλογέ για μια χώρα σαν το ε, για μια χώρα που κατά το ίμιση μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί. Και έχουμε επίση κάποιε περιοχέ όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμεί αλλά και η κυβέρνηση περισσότερα, να βελτιώσουμε δηλαδή τις εκλογικές λειτουργίες και διαδικασίε και ένα από τα βασικό λάθο ήταν ότι μετά τις εκλογές του 4 και του 5 διαλύθηκε ο μηχανισμός, ο εκλογικός. Οπότε αρχίσαμε από το Α. Ιδίω όσον αφορά την Επιτροπή των Καταγγελιών και αυτή εξ αρχή υπήρξε θέμα ε, του κατά πόσο η εκλογική επιτροπή ε, ήταν ε, ανεξάρτητη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά το πώς συμπεριφέρθηκε αυτό το όργανο μετά. Και αυτή η ανεξάρτητη εκλογική επιτροπή θεωρήθηκε ότι καθόλου η εκλογική διαδικασία δεν ήταν αμερόληπτη. Και επίσης ε, υπήρχαν προβλήματα και στους εκλογικούς καταλόγους. Κάποια εκατομμύρια πολιτών ε, έλαβαν ειδοποίηση να ψηφίσουν ενώ δεν δικαιούνται. Και αυτό φυσικά είναι στοιχείο νοθείας. Επίσης κάτι το οποίο δεν φροντίσαμε ήταν ε, η ασφαλής συμμετοχή των γυναικών στι εκλογέ. Φυσικά και ανέκυψε, αυτή, η, ανέκυψε αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ αργά. Πολύ αργά η διεθνή κοινότητα άρχισε να ε, προσέχει το τι γίνεται στα εκλογικά κέντρα των γυναικών. Τελευταία στιγμή βρέθηκε κάποιος ειδικό σύμβουλος, για παράδειγμα. Όλα αυτά βεβαίω αποξένωσαν τις γυναίκες από τις εκλογές, απέσχουν. κάτι το οποίο επίσης συνέβαλε στο να έχουμε σε πολλές περιοχές της χώρας. Ελπίζουμε στο μέλλον να, να μην επανελθούν αυτά τα λάθη, γιατί του χρόνου έχουμε γεωλογικές εκλογές και άρα ελπίζουμε να έχουμε καλύτερες επιδόσεις τότε. Να λυθούν τα προβλήματα εκλογικών καταλόγων, ε, τα προβλήματα της ε, αμεροληψίας των εκλογικών ε, φορέων, οργανωτικών φορέων, συμμετοχή των γυναικών. Επίσης, οι ενστάσεις είναι πάρα πολύ περιορισμένες οι ρυθμίσεις για τους ε, υποψηφίους και για κάθε του ένσταση και τελικά ούτε εδώ βοηθήσαμε Ούτε εδώ δεν διαπιστώθηκε κατά πόσο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ένσταση κατά υποψηφίων. Άρα ελπίζουμε στο μέλλον να τα καταφέρουμε καλύτερα. Ιδάλω θα καταλήξουμε σε ένα κοινοβούλιο στη χώρα που θα έχει για βουλευτές τους πολέμαρχους, τους απατεώνες και εγκληματίες. Πάντω, τώρα η διεθνή κοινότητα έστειλε τη μεγαλύτερη ε, δυνατή επιτροπή παρατηρητών, ομάδα παρατηρητών. Έχει συνταγή μια πρώτη έκθεση. Η ανακοινώσει τύπου στην αρχή τα είπαν τα πράγματα πολύ πιο ρόδινα και όσον αφορά αυτή την νοθεία, τη βία και την αποχή, τα σχετικά προβλήματα αλλά και σε σχέση με τις δυνατότητες που είχαν οι παρατηρητές να κάνουν τα καθήκοντά τους, να τα ασκήσουν. Όλα αυτά θα φυγούν σε αυτήν την έκθεση, την τελική της μορφή, που ελπίζω να τα λέει λιγότερο ρόδινα. Ούτως ώστε να ξαναβρει η χώρα την αξιοπιστία της και η διεθνής κοινότητα. και οι ίδιοι οι παρατηρητές μας διακυβεύουν την αξιοπιστία τους σε αυτά που θα έχει έκθεση. Τώρα για τα δικαιώματα των γυναικών. Κάποιο νομοσχέδιο εγκρίθηκε την άνοιξη, Εγκρίνεται η αποχώρηση των γυναικών από το σπίτι, η αναχώρηση χωρίς προηγούμενη έγκριση. Όλα αυτά ήταν κατόπιν κάποιες διεθνούς κατακραυγές. Υπήρξε μεγάλη πίεση προς τον πρόεδρο της χώρας για να προβήσει αναθεώρηση του σχετικού δικαίου της χώρας. Πέρασε λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο. Ε, μετά ανεκλήθησαν κάποιες από αυτές τις διατάξεις, αυτό έγινε μέσω των εκλογών, τόσο ώστε να μπορέσει να ε, αποσπάσει κάποιες ε, ψήφους κάποιων ε, ακραίων θρησκευτικών στοιχείων, σιητών και διεθνής κοινότητα δεν είπε τίποτα. Αυτό είναι επομένω για του φονταμεταλιστέ. Αυτό όμω φυσικά και θα έχει επιπτώσει όσον αφορά τα βήματα πρώτα που έχουν προηγουμένω σημειωθεί όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Άρα θα πρέπει και σε αυτά τα θέματα να παρέμβει η διεθνής κοινότητα γιατί είδαμε ότι αποδίδει η πίεση όταν ασκείται τώρα. Είχαμε προεδρικό διάταγμα τον Ιούλιο ε, σε σχέση με τη βία κατά των γυναικών, το οποίο όμως ακόμα δεν έχει γίνει νόμος του κράτους. Αυτό είναι μια μικρή ε, βελτίωση τα δικαιώματα των γυναικών. Φύγεται και για πρώτη φορά το έγκλημα του βιασμού. Όμως, χρειάζεται και εδώ να τους βοηθήσουμε ε, τεχνική αερογή, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει πράξη αυτή η ιδέα, αυτό το διάταγμα. Ένα τελευταίο θέμα για τα δικαιώματα των γυναικών. Όλα είναι και περισσότερο στηρίζεται η κυβέρνηση στα συντηρητικά στρώματα του πληθυσμού και έγινε συζήτηση όσον αφορά τι επαφέ και διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν, γιατί προ τα εκεί πηγαίνουμε. Και θεωρούν σαν στρατηγική εξόδο από το διέξοδο όλων των εμπλεκομένων χωρών το να έρθουν σε επαφή με τους Ταλιμπάν. Δεν θα το σχολιάσω, θεωρείται από τους, πολλού πολλούς ότι αυτό είναι η μοναδική διέξοδο στο διέξοδο. Όμως, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα δικαιώματα των γυναικών σημαίνει πολλά αυτή η ε, σύγκληση με τους ε, τέλους. Όταν ε, κλείνονται τα πολιτικά deal, φυσικά και έχει αποδειχθεί ότι δεν πληρώνονται τα δικαιώματα των γυναικών τώρα όσον αφορά την αντιμορρυσία. Όλα αυτά που λέμε αλληλοσυνδεδεμένα είναι. Όμως, αυτή τη στιγμή, όσο πέραν γύρω από τις εκλογές, βλέπουμε ότι θα ασκηθεί κάποια επιρροή στη σύνθεση και πολιτική της επόμενης κυβέρνησης από τις εκλογές. Η κυβέρνηση ήδη έχει κάνει κάποια έχει κλείσει κάποιες συμφωνίες με κάποιους πολέμαρχους, έχουν δοθεί πάρα πολλές ε, υποσχέσεις να τους δώσουν δουλειά και όταν τελικά κατακάτσει ο κουρνιαχτός των εκλογών θα έχουμε εξελίξεις και μας προβληματίζει το ότι δεν υπάρχει κανένας είδους ε, μηχανισμός προβολής ενστάσεων. Θα πρέπει όμως το σύστημα να ισχυροποιηθεί να βοηθήσει τη διεθνή κοινότητα όσον αφορά το capacity building, όσον αφορά την, τη στελέχωση του μηχανισμού, του κρατικού και θα έπρεπε οι διορισμοί των υπαλλήλων να είναι περισσότερο εξωκρατικοί διότι διαπιστώνουμε ότι συνεχίζονται οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων ε, σε μια χώρα που εγκληματίες, πολέμαρχοι ε, ουσιαστικά έχουν ανοιχτού του διάβλους της εξουσίας και κινούνται υπεράνω του νόμου. Πολιτική πίεση χρειάζεται και σοβαρότερη αντιμετώπιση. Να προσπαθήσουμε να πιέσουμε μέσω της οικονομικής βοήθειας, μέσω των όσων δρούν και επενδύουν στο Αφγανιστάν. Γιατί αλλιώς δεν θα προχωρήσει καθόλου η υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα me Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε με πολύ προσοχή όλη την ε, σημασία των δικαιωμάτων της γυναίκας σε αυτή τη συζήτηση και σε αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης των εκλογών. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα που έχουν οι γυναίκες πλέον να συμμετέχουν στις εκλογές. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε πάντοτε υπόψη. Σας ευχαριστούμε πάντως που αναφέρατε επίσης αυτό τον νόμο που ε, διακρίνει τις γυναίκες και που μάλλον που αποτελεί διάκριση εναντίον των γυναικών και που είναι ενάντιος στα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν αρκεί δηλαδή να έχει κανείς ένα σύνταγμα ώστε να τηρούνται τα γυναικεία δικαιώματα. Θα πρέπει να μην υπάρχουν τέτοιου είδους νόμοι. Εν πάση περιπτώσει αυτές οι πληροφορίες είναι όλες εξαιρετικά πολύτιμες για μας που χρέο έχουμε να μεριμνήσουμε για την χρήση αυτών των, ε, των οικονομικών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με αυτήν την εκλογική διαδικασία. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση και ποιες είναι οι συνέπειες των όσων συνέβησαν. Και τώρα στρέφομαι προς τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, έχετε κάποια λεπτά στη διάθεσή σας για να μας εξηγήσετε ποια είναι η κατάσταση και να μας εξηγήσετε και ποια είναι η θέση του, της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας πως είναι πολύ καλό που έχουμε τον κύριο Λάγκερ εδώ που μας έχει έρθει από την Καμπούλ. Εμείς παρακολουθούμε στενά την δουλειά που κάνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αφγανιστάν και ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά της γιατί πρέπει ε, καταρχήν να συνδυάσει το ρόλο της ως κυβερνητικός θεσμός ενώ προσπαθεί να προωθήσει το σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεων ε, του Αφγανιστάν πράγμα το οποίο υποστηρίζει βέβαια και η διεθνή κοινότητα. Επίσης, συμφωνούμε με μέγα τμήμα της ανάλυσης που ακούσαμε. Μου θυμίζει, πρόεδρε, αν δεν ξέρω αν το είδατε, την γελιογραφία στη χθεσινή International Herald Tribune που λέει ο Μποάμα στον Καζάη «Δεν καταλαβαίνεις τη δημοκρατία» και ο πρόεδρος Καζάη απαντά «Εσύ δεν καταλαβαίνεις το Αφγανιστάν». Περιέχει ένα τμήμα αλήθεια σε αυτή η γελιογραφία. Εμείς Ανέκαθεν πιστεύαμε και προσπαθούσαμε να πείσουμε τους Αυγανούς συναδέλφους να προχωρήσουν επικυρώνοντας τους βασικές συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να αναπτύξουν τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Και όντως έχει γίνει μεγάλη προ... πρόοδος, είναι μεγάλη διαφορά από τις ημέρες των Ταλιμπάν. Ε, ωστόσο είναι ακόμα αλήθεια ότι μπορεί κανεί να επικυρώσει μια συνθήκη, αλλά καταρχήν πρέπει να εσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία και έπειτα πρέπει και να εφαρμοστεί. Και έχουμε δει ότι η ελευθερία λόγου και ΜΜΕ έχει υποστεί πιέσει τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό το λόγο η Ένωση μαζί με την Ορβηγία εξέδωσε μία δήλωση για την ελευθερία των ΜΜΕ φέτος. Να σας προσθέσω ότι ανησυχούμε πολύ γιατί η κατάσταση των γυναικών έχει όντως επιδεινωθεί από ορισμένες απόψεις και θα επανέλθω σε αυτό. Το βασικό μας θέμα βέβαια είναι αυτό των εκλογών. Αυτές ήταν οι πρώτες εκλογές που έγιναν από ε, την Αφγανική καθοδήγηση και υπήρχε βέβαια η επιδεινόμενη κατάσταση ασφαλείας ε, ε, και η ένταση με το Ιράν και αυτό ήταν ήδη μεγάλη πρόκληση υπάρχουν κάποια τμήματα της χώρας όπου η προσέλευση στις εκλογές ήταν εξαιρετικά χαμηλή. Νομίζω στο Κανταχάρ ήταν λιγότερο από 10%. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία μέσω της ε, πιστολής παρατήρησης της οποίας ηγήθηκε ο στρατηγός Μοριών και βρισκόταν βρίσκεται από τον Ιούλιο εκεί και πρέπει να παρακολουθήσει τις εκλογές, ε, τα θεσμικά όργανα σε και τη χώρα και ελπίζουμε ότι θα μας δώσει κάποια αποφθέγματα, κάποια δάγματα καθώς προχωράει η εκλογική διαδικασία και όπως σωστά και τονίστηκε μετά από τις προεδρικές εκλογές τώρα πρέπει να δούμε και τις κοινοβουλευτικές εκλογές που θα πρέπει να γίνουν πριν από τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Θα είδατε ότι οι αποστολές παρατήρησης των εκλογών δήλωσαν τη στιγμή των εκλογών κάποια πράγματα που ε, μάλιστα συμπληρώθηκαν από μια περαιτέρω δήλωση για το γεγονός ότι το έργο τους επιδεινώθηκε και ε, περιπλάκει λόγω του ότι η ανεξάρτητη Επιτροπή για τις εκλογές επέλεξε να εκδώσει αρχικά τελικά αποτελέσματα δίνοντας στον κύριο Καζάη πάνω από το 50%. Μάλλον για να αποφευθεί μια, ένας δεύτερος γύρος. Ε, αυτό κάποια στιγμή όπου υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα για το ποια ακριβώς στοιχεία συμπεριλαμβάνονταν σε αυτό το σύνολο που δόθηκε στη δημοσιότητα και υπάρχουν ε, παράπονα νομίζω 2.200 200 καταγγελίες οι οποίες ακόμα διερευνώνται. Γύρω στους 600 εκλογικά γραφεία θεωρούνται ύποπτα. Ορισμένα θεωρούνται ως εκλογικά γραφεία ε, φαντάσματα. Τώρα, αν ε, τα υποθεμένα αποτελέσματα βρίσκονται στο σύνολο ή όχι, δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι αλλά πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που η διαδικασία αυτή έγινε, που το IEC και η Εκλογική Επιτροπή Καταγγελιών αναλαμβάνουν πλήρων τις ευθύνες τους. Το να προκαταβάλουμε τις αποφάσεις τους ακριβώ θα σήμαινε να ζημιώσουμε αυτά τα θεσμικά όργανα, των οποίων εξοπιστή είναι πολύ σημαντικά για την δημογραφική ανάπτυξη του ναι. Αφγανιστάν. Στο ίδιο πνεύμα, η η αποστολή παρατήρησης των εκλογών είναι εκεί και θα παραμείνει επιτόπου μέχρι ότου ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία, μέχρι ότου αποφασιστεί να θα γίνει ή όχι δεύτερος γύρος, θα βρίσκονται εκεί και μόνο τότε θα μπορέσουμε επί τη βάση της πλήρους εικόνας να συντάξουμε μια πλήρη έκθεση για τη διεξαγωγή των, προ... προεδρικών εκλογών του Αφγανιστάν και να εκδώσουμε και τις πρακτικές συστάσεις που σας ανέφερα. Όπως υπόθηκε, η προετοιμασία των εκλογών του επόμενου έτους είναι επίσης προτεραιότητα, διότι πιθανά υπάρχουν, είναι ακόμα πιο σημαντικό να ενισχυθεί ένα δημοκρατικό σύστημα και εν γέννη μια δημοκρατική κυβέρνηση στο Αφγανιστάν. Και γι' αυτό και πιστεύω, ελπίζω μάλλον, θα υπάρξει μια δυνατότητα για επαφές με τη νέα κυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα, ώστε οι συστάσεις μας να ακολουθηθούν. Μια διαδικασία, μάλλον συζήτηση, τώρα για την επόμενη, για την συνεχιζόμενη διαδικασία Θα πρέπει αυτό να συνδεθεί με την αφοπλισμό των παράνομων ομάδων. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι πως δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Θα πρέπει να χειριστούμε τα θέματα αυτά και είναι σαφές πως οι κοινοβουλευτικές εκλογέ θα είναι μια πραγματική δοκιμασία. Um, Το θέμα της ε, μετάβασης ε, στην δικαιοσύνη είναι επίσης πολύ δύσκολο θέμα μέσα στο σημερινό πολιτικό πλαίσιο, αλλά είναι απαραίτητο για την νομιμότητα της κυβέρνησης. Διότι οι εκπρόσωποι τη είτε στο κοινοβούλιο είτε σε δημόσια λειτουργήματα θα πρέπει να είναι υπόλογοι ε, και να λογοδοτούν για παρελθούσες και μελλοντικές τους ενέργειες. Ας δούμε τώρα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα γνωρίζετε πιθανότατα ότι το Συμβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν και από τη Γραμματεία του Συμβουλίου να εξετάσει μια νέα προσέγγιση προς το Αφγανιστάν αλλά και προς το Πακιστάν ε, παρεπιπτόντως και αυτό α, μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Ελπίζω πως αυτό θα καταλήξει σε ένα έγγραφο που θα δίνει πολύ μεγαλύτερη έμφαση για, τα πρότυπα πολιτικής συμπεριφοράς είτε επανεπιβεβαιώνοντας το κράτος δικαίου στην συνταγματικότητα των κυβερνητικών ενεργειών, είτε μειώνοντας το επίπεδο διαφθοράς, είτε κάνοντας ε, κάτι για να υπερασπιστεί τα, τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό αν θέλουμε πραγματικά επιτυχώς να συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση αλλά είναι σαφές εδώ και χρόνο, εδώ και καιρό, ότι θα είναι πολύ δύσκολο να εγκαθιδρύσει μια κάποια αξιοπιστία απέναντι στο λαό του, είτε μιλάμε για ασφάλεια, είτε για τη διοίκηση των επαρχιών, είτε για την παροχή των υπηρεσιών και όχι βέβαια λιγότερο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά των γυναικών. Το γεγονός ότι τελευταία στιγμή πέρασε από την μεταβατική κυβέρνηση η νομοθεσία η θρησκευτική για τις γυναίκες δεν καθιστά ευκολότερο το έργο αυτό για την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Επίσης, βία κατά των γυναικών και ο σχετικός νόμος ήδη είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες και τη στιγμή που η έκθεση του ΙΕ δείχνει ότι αυξάνεται η βία κατά των γυναικών, ιδιαίτερα των γυναικών που είναι δημόσια πρόσωπα. Ακόμη πιο προβληματικό είναι ένα γενικό πρόβλημα στο Αφγανιστάν και αυτό είναι η καταλληλότητα του δικαστικού συστήματος ώστε να υπάρξει μια πραγματική ποινή Τέλος, δεν επιβεβαιώνεται ούτε η ανεξαρτησία του εθνικού αναμεταδότη του Άρθια, γιατί το Κοινοβούλιο είπε ότι θα έπρεπε να οριστεί, να διοριστεί από τον πρόεδρο ο διευθυντής ε, του σταθμού αυτού. Εμείς το θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα όσον αφορά τα στάνταρ, τα πρότυπα της πολιτικής ζωής του Αφγανιστάν. Kiitos erittäin paljon komission edustajalle. Nyt on kuitenkin aika suorasanaisesti sanottava, että, että parlamentin näkökulmasta Ευχαριστώ. Για να δούμε και την άποψη του Κοινοβουλίου για τις εκλογές αυτές. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε προκειμένου ότι οι βασικές συνθήκες για τη διαδικασία αυτή, την εκλογική αυτή διαδικασία, δεν τηρήθηκαν. Μας εξήγησε βέβαια η Επιτροπή ποια ήταν η κατάσταση. Λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα δεδομένα. Ας ακούσουμε λοιπόν τους συναδέλφους που θέλουν να λάβουν το λόγο. Να σας διαβάσω και τον κατάλογο. Θέλει κι άλλος το λόγο. Ναι, βεβαίως, να σας καταγράψω και εσάς. Αφού είναι τόσο πολλοί λοιπόν οι συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο, Παρακαλώ να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι για να ακούσουμε και τις απαντήσεις των προσκεκλημένων μας. Η κυρία Αντρέκη, Κινέ, Αντιπρόεδρος. Πρόεδρε, ευχαριστώ και δεν ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι έλαβαν το λόγο για τις παρεμβάσεις τους. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Πριν από ένα χρόνο περίπου είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το Αφγανιστάν. Συναντηθήκα με υπουργούς της κυβέρνησης στην Καμπούλα ε, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και την επαρχία του Γκόρ ε, που μίλησα με τον κυβερνήτη και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Όλοι ήδη μιλούσαν για τις εκλογές και μίλησα και με εκείνους που κανονικά ασχολούνται με την ε, προπαρασκευή της εκλογικής διαδικασίας. Και με ενδιαφέρον τώρα παρακολουθώ την έκβαση αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Για τον κύριο Λάγκαρη. Ο Φιλίπ Μοριγιόν, επικεφαλής της ομάδας ε, παρατηρητών των εκλογών, έκανε μετά τις εκλογές την εξή δήλωση και παραθέτω. Παρατηρήσαμε μια μεθοδολογία εκλογική καλή, ισότιμη, δίκαιη, αλλά δεν ήταν ελεύθερες εκλογές λόγω της τρομοκρατίας που επικρατούσε σε αρκετές περιοχές. Ερωτώ λοιπόν εάν συμφωνείτε με την εκτίμηση αυτή του κυρίου Μοριγιόν. Και η ερώτηση προς όλους τους ομιλητές τι θέση έχετε, τι ανάλυση κάνετε της παρουσίας των διεθνών παρατηρητών στις εκλογές. Ήταν ικανοποιητική η παρουσία τους επαρκής. Επίσης, εάν υπάρξει άλλος ένας γύρος εκλογών, δεν υπάρχει ο κίνδυνος οι Ταλιμπάν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή για ακόμη περισσότερη τρομοκρατία. Εχθές από κάποιο διεθνές κανάλι παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου του επικεφαλής της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος είπε ότι θα χρειαστούν δύο-τρεις μήνες τουλάχιστον για να διερευνηθούν όλες οι ενστάσεις. Πράγμα το οποίο ασφαλώς θα φέρει ακόμη περισσότερη αστάθεια στη χώρα. Για τη συμμετοχή των γυναικών δεν διατυπώνω ερώτηση, το καλύψατε όλοι το θέμα αυτό, αλλά ασφαλώς πολλά θέματα έχουν να συζητηθούν στο ε, ζήτημα αυτό. Αλλά για να κερδίσουμε χρόνο. Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν ικανοποιητική. Ήταν ισότιμη, ήταν αμερόληπτη. Όταν είπατε ότι για ένα λεπτό παρουσία στην τηλεόραση ένας υποψήφιος έπρεπε να καταβάλει 600 δολάρια, προφανώς δεν μπορούσε κανείς δωρεάν να εξασφαλίσει χρόνο τηλεοπτικό. στα αγγλικά. Είμαι υποχρεωμένη να σημειώσω το δυσάρεστο, να κάνω τη δυσάρεστη παρατήρηση ότι ε, εάν όλοι έχουν τόσο πολλές ερωτήσεις όπως η Αντιπροέδρος δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε ποτέ. Η κυρία Μενρόιτσεν. Εγώ θα είμαι σύντομη Πρόεδρε. Και ευχαριστώντας τους ομιλητές θα ήθελα να διατυπώσω το εξής ερώτημα. Ακούσαμε τόσο είπατε. Για τους παρατηρητές και δεν θέλω να μου πείτε τι γνώμη διατύπωσαν εκείνοι γιατί έχω την εντύπωση ότι τι πρώτες μέρες μετά τις εκλογές ήταν πολύ πιο θετικά τα σχόλιά τους από ό,τι διαπιστώσαμε στην συνέχεια. Ε, και γι' αυτό ερωτώ, γιατί αυτή η απόκληση ε, πρόβλημα οργανωτικό, Ενδεχομένω, ήρθαν περισσότερα στοιχεία κτλ. Και δεύτερον, τι διδάγματα αντλείται από το γεγονός αυτό και από τις εκλογές βέβαια για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Επίσης για τις γυναίκες, ξέρουμε ότι η κατάσταση των γυναικών, των ε, δικαιωμάτων της γυναίκας δεν είναι ικανοποιητική εκεί. Και ρωτώ τι πιστεύετε ότι μπορεί να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος Χάουιτ, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Και στο συγγνώμη από τον Επίτροπο, γιατί άργησα να φτάσω και δεν άκουσα όλη την παρέμβαση. Αλλά είχα πάει και εγώ όπως ε, και αντιπρόεδρος στο Αφγανιστάν. Με ε, α, ενδιαφέρον άκουσα τόσο είπατε. Και το ότι είναι πιθανόν να βοήθησε η παρουσία των ε, παρατηρητών στην ε, εκλογική διαδικασία. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι βέβαια οι παρατηρητές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι τα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι μπορείτε εσείς στο Αφγανιστάν να αξιοποιήσετε την παρουσία τους εκεί και να βελτιώσετε την κατάσταση. Και επίση για την Επιτροπή των Εξωτερικών, θέλω να πω ότι θα ήταν χρήσιμο να δούμε τον στρατηγό Μοριό όταν επιστρέψει από την αποστολή του εκεί για να μα μιλήσει από πρώτο χέρι. Επίση, ε, για το θέμα των εκλογών και των παρατηρητών, ε, θα ήθελα να σημειώσω ότι έχουμε, αν όχι από το Αφγανιστάν, πάντως από άλλες χώρες, πολλές ε, αποστολές στο παρελθόν ε, όπου σημειώθηκαν προβλήματα, παρατυπίες ε, σε διάφορα σημεία. Και αυτό που εξασφάλισε την πρόοδο ήταν το ότι ε, εισακούστηκαν οι παρατηρήσεις των παρατηρητών αυτών και διορθώθηκαν τα προβλήματα. Ο Καρζάη με τα ποσοστά που έχει εξασφαλίσει πιστεύετε ότι μπορεί να στηριχθεί στην υποστήριξη του λαού ή όχι εάν δεν επαναληφθεί η διαδικασία. Επίσης, πιστεύετε ότι οι παρατυπίες που έλαβαν χώρα ήταν μια οργανωμένη προσπάθεια για ενώθευση των εκλογών, για ανατροπή του αποτελέσματος ή ήταν απλώς φαινόμενο που προκάλεσε η αστάθεια, η ανασφάλεια, οι δύσκολες συνθήκες στις οποίες εξήγησαν οι εκλογές. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι δεν ε, βρίσκω χρήσιμο το να λέει κανεί, ε, όπω άκουσα, να βελτιωθούν οι διαδικασίε την επόμενη φορά και να προσέξουμε τελικά. Φυσικά και πρέπει να γίνει αυτό, αλλά δεν αρκεί. Τώρα πρέπει να δούμε τι γίνεται και δεν ε, κάνουμε τίποτα εμείς στις Βρυξέλλες να σταυρώσουμε τα χέρια και περιμένουμε την επόμενη εκλογική διαδικασία για να δούμε αν υπάρχουν άλλα προβλήματα και άλλη νοθεία. Δεν έχουμε χρόνο λοιπόν, θα είμαι σύντομο. Αλλά παρακαλώ την Επιτροπή, το Human Rights Watch να μας πει τι παρατηρήσεις έχει ως προς την τήρηση των ε, διαδικασιών. Και επίσης για όλους τους ομιλητές ο Ομπάμα, ο Μπράουν και άλλοι, από ό,τι φαίνεται, επισημαίνουν ότι θα γίνουν προσπάθειες για ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν. Εν ώψη της κατάστασης που προκύπτει. Βέβαια δεν μπορώ να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι θα τα καταφέρουν, αν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ασφάλειας, αλλά αυτό που μπορώ να ρωτήσω εσάς είναι εάν θεωρείτε ότι είναι σε θέση αυτές οι δυνάμεις ασφαλείας να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Εθνικό ανθρωπιστικό δίκαιο. Ή σε ποιο βαθμό μπορούμε να περιμένουμε κάποια ανεξέλιξη και πρόοδο στο μέλλον. Κύριε Χάρη, του ευχαριστούμε. Κύριε Κασάκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα με να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας διότι μας ε, ενημέρωσαν πάρα πολύ καλά έτσι αποδεικνύεται ότι το Αφγανιστάν είναι όντως μία από τις πιο φτωχές χώρες και ότι ο λαός έχει υποφέρει πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες. κατά πάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχής πόλεμη ε, Το βιωτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό και θα πρέπει με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο να ρωτήσω κάτι τους προσκεκλημένους μας πρώτα πρώτα όσον αφορά το των εκλογών. Ακούσαμε τους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανισμών αλλά ε, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουμε μια σειρά παραβάσεων που έλαβαν χώρα. Τι σημαίνει αυτό. Τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Τι επίδραση θα έχουν αυτές οι εκλογές τις επόμενες. Τι θα κάνουν αυτοί οι οποίοι εξελέγησαν στην διεθνή σκηνή. Τώρα, όσον αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας. είδα μια ταινία. Ήταν η ιστορία μιας κοπέλας που είχαν υποχρεωθεί οι γονείς της να την ε, μεταμφιάσουν σε άντρα για να την προστατεύσουν από τους Ταλιμπάν, ούτως ώστε να μπορεί να πηγαίνει σχολείο. Όμως, τελικά ξεσκεπάστηκε. Και πέφερε πάρα πολύ μετά. Τι πιστεύετε όσον αφορά τη νέα νομοθεσία για τις γυναίκες. Θεωρείτε ότι είναι επαρκής. Το Αφγανιστάν έχει προσχωρήσει μια σειρά διεθνών ε, συνθήκων που κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα συνεχίσει η χώρα να τηρεί τις υποχρεώσεις της, της διεθνής. Ευχαριστούμε κύριε Καζάκ. Και αυτός ο κύκλος ερωταπαντήσεων θα κλείσει ε, με την Σβένσον, η οποία θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή των ε, Γυναικείων Θεμάτων. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε ε, στη σημερινή συνάντηση. Όπως ε, λέχθη, συμμετέχω στην Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών. Ελπίζουμε ότι θα είναι εργαστή η συνεργασία με την δική σα υποπιτροπή, κυρία Πρόεδρε. Γιατί άλλωστε είναι κοινό αγώνα των ανθρωπίνων, των δικαιωμάτων τη Γυναίκα. Άκουσα και ευχαριστώ όλου τους εσμηνού μα συγητές. Έχω κάποιε παρατηρήσει και ερωτήσει. μια που πρώτα πρώτα στην αρχή της ε, παρέμβασης της κοινότητας στο Αφγανιστάν ξεκίνησε αυτός ο αγώνας για την κατοχή ε, κατοχήρωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου όμως παρότι πέρασαν τόσα χρόνια ε, έχουν μάλλον παραμεληθεί τα δικαιώματα αυτά και ο αγώνας για την κατοχήρωσή τους θεωρώ ότι αυτό έγινε γιατί πρώτα πρώτα η διεθνή κοινότητα για πολύ καιρό μάλλον αφελώς αντιμετώπιζε την ε, καταπίεση της γυναίκας στο Αφγανιστάν και επομένως παρά όλη την καλή θέληση καθέστηκε δύνατο να βοηθήσουμε από κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ε, πλευράς της γυναίκας στο Αφγανιστάν. Ε, η ένοπλη αντιπαράθεση έβαλε στο περιθώριο το πρόβλημα του δικαιωμάτων της γυναίκας. Δεν θεωρήθηκε θέμα πολιτικά σημαντικό, θέμα ασφάλειας, ε, υπόθεση της γυναίκας μέσα σε αυτές τις συγκρούσεις. Άρα, στα πλαίσια τη θετική μα για τη χώρα αυτή να προσδώσουν περισσότερη σημασία στο γυναικείο ζήτημα. Μπορεί να βοηθήσουν οι γυναίκε στην εξομάλυνση τη κατάσταση στη χώρα. που στηρίζουν την οικογένεια, οι κοινότητε που πλήσονται άμεσα από τι συγκρούσει εκεί. Μπορούν να ωφεληθούν. Και όσον αφορά τώρα τις εκλογές και τις συμμετοχές εκλογές, είχαμε φοβισμένους πολίτες, καταπιεσμένους πολίτες που δεν μπόρεσαν βέβαια να ψηφίσουν ή και να ψήφισαν δεν ψήφισαν ανεξάρτητα. Αυτό ισχύει φυσικά και για γυναίκες και για άντρες. Και επί τη βάση στοιχείων που έχω, γνωρίζω ότι είχαμε να στον αφορά τους εκλογικούς καταλόγους των γυναικών. Υπήρξε κάποιο επιλογή δικαίωμα επιλογή τη γυναίκα, αν θέλει να ψηφίσει ή όχι. Οπότε και γι' αυτό το λόγο είχαμε ενωθεία με δημιουργία ψηφοφόρων φαντασμάτων. Γυναικών ψηφοφόρων που δεν υπήρχαν. Πότε σας παρακαλώ ενημερώστε με. Ε, έτσι έχει κατάσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε. Και επαναλαμβάνω, ελπίζω ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία ε, υπό Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Επιτροπή των Δικαιωμάτων τη Γυναίκα. γιατί είναι κοινά τα συμφέροντα, κοινό αγώνα από πολλέ απόψει. Ευχαριστώ και πάλι. Kiitos rouva Svensson. On aivan selvää, että ihmisoikeus alivaliokunnalla ja teidän johtamallanne naisten oikeus. Πρόεδρος. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και εμείς βέβαια πώς και πώς περιμένουμε το πώς θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή σας, υπό την Προεδρία σας. Προσοχή μου στα, χρονικά πλαίσια, ο Μπιόλς Νίλσον, Τσίπ, θα μου το λόγο. Και μετά θα δώσουν τις απαντήσεις οι, okay, προσκεκλημένοι μας. Πρώτα πρώτα επομένως απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους τρεις μας προσκεκλημένους. Very serious question also. Πολύ σοβαρή μια μεγάλη σειρά ερωτήσεων, δύσκολες ερωτήσεις σε σχέση με την ημερομηνία των εκλογών και το ρόλο των διεθνών παρατηρητών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω μαζί μου, 1.106 διεθνείς παρατηρητές από 50 διεθνείς οργανισμούς συμμετείχαν στην πλήρη παρατήρηση των εκλογών. Αλλά εφόσον η ασφάλεια ήταν πολύ άσχημη σε εκείνη τη μέρα, ακόμα και στην Καμπούλ εκείνη την ημέρα, δεν υπήρχε κυκλοφορία, δεν υπήρχε συμφόρηση. Πολλοί κόσμος φοβήθηκε και έμεινε σπίτι του. Η οικογένειά μου, για παράδειγμα, πήγε σε ένα πολύ κοντινό εκλογικό κέντρο και γύρισε πίσω πάρα πολύ σύντομα και Πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης επίσης και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ανέπτυξε 300 ανθρώπους σε ολόκληρο το Αφγανιστάν δεν είδε καθόλου παρατηρητές, διεθνείς παρατηρητές σε, στα εκλογικά κέντρα. Λόγω των δύσκολων προβλημάτων ασφαλείας. Δεν έχω ωστόσο λεπτομέρειες για το πού βρίσκονταν. Πάση περιπτώσει αφού ήρθαν στο Αφγανιστάν και έκαναν ανακοίνωση τύπου και πίεσαν τα πράγματα, αυτό ήδη εκτιμήθηκε. Είχαμε και αρκετού παρατηρητέ από ασιατικέ χώρε καθώ και Ευρωπαίου. Now, how to do with this. Η υπόθεση τώρα, η κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Όσοι έχουν ε, ταξιδέψει λίγο στο Αφγανιστάν θα γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση των γυναικών. Το πρόβλημα δεν είναι να τους μάθουμε μόνο να γράφουν και να διαβάζουν. Το πρόβλημα είναι να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική κατάσταση. Ακόμα και την ημέρα των εκλογών, πολλές γυναίκες δεν αναγνώριζαν καν τις εικόνες των υποψηφίων και δεν μπορούσαν να διαβάσουν τον αριθμό το κάθε υποψηφίου. Ποιος είναι ο 35ος, ποιος είναι ο 36ος και το καθεξής. Και οι σύζυγοί τους, οι άλλοι, τους έδειξαν ότι έπρεπε να ψηφίσουν για το ΔΑΔΕ, το ΔΙΝΑ. Αν κανείς βγει από την Καμπούλ θα δει πόσο άσχημη είναι η κατάσταση των γυναικών. Χρειάζεται μεγάλη υπομονή και προσπάθεια για να βελτιωθεί η κατάστασή τους, ώστε να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να βελτιώσουν την κατάστασή τους. Να απαιτήσουν για τον εαυτό τους. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες, λίγες, που είναι δραστήριες στο κοινοβούλιο, Αυτό είναι πολύτιμο, αλλά σε σχέση με όλες τις γυναίκες του Αφγανιστάν πρέπει να πω ότι είμαστε σε πρωταρχικό στάδιο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Υπήρξε μια ερώτηση ενός συναδέλφου όσον αφορά τις δυνάμεις ασφαλείας, για το πώς δηλαδή αυτές μπορούν να βελτιωθούν. Αυτό παίρνει πολύ καιρό δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Εθνικό Στρατό και στην Εθνική Αστυνομία. Νομίζω πως ακόμα και αν αύριο οι διεθνείς δυνάμεις ανακοίνωναν πως τα μαζεύουμε αύριο και φεύγουμε μετά από δύο-τρεις μήνες έστω και ένα χρόνο, θα γινόταν μια μοιρασιά ανάμεσα στο στρατό και την Εθνική Αστυνομία για το πώς θα μοιράσουν την τη χώρα. Και εκείνη την ημέρα, την επόμενη μέρα που θα φεύγαν οι διεθνείς δυνάμεις, η Καμπούλ θα χωριζόταν σε κομμάτια για το ποιος θα διοικεί πού. Χρειάζεται λοιπόν η παρουσία των διεθνών δυνάμεων. Και πριν από μερικέ μέρε, οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί ανακοίνωσαν ότι θα παραμείνουν στο Αφγανιστάν για πιο μακρά περίοδο, εκτό αν είναι βέβαιοι πω ο Εθνικό Στρατό και η Εθνική Αστυνομία ήταν σε θέση να δυσφαλίσουν το Αφγανιστάν. Αυτό είναι πολύτιμο για μας. Και αυτή η ανακοίνωση πιστεύω πως ε, έχει, βάλει σε, έχει υπογοητεύσει τους Ταλιμπάν γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν. Όσον αφορά τις διεθνείς δυνάμεις, εκφράζουν την ανησυχία τους, την απογοήτευσή τους με τον ίδιο τρόπο που οι Ταλιμπάν ανησυχούνται. Καλύτερος τρόπος είναι λοιπόν να προκαλέσει κανείς τους Ταλιμπάν από τη διεθνή κοινότητα ότι δηλαδή να δείξει η διεθνή κοινότητα είναι σοβαρή απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Το Αφγανιστάν απέτυχε με τους Ταλιμπάν. Ο εκπρόσωπος τη Κομισιόν ανέφερε μια γελιογραφία που ο Ομπάμα λέει ότι δεν ξέρει, δεν, στον Καρζάι ότι δεν ξέρει τη δημοκρατία και ο άλλο απαντά μα εσύ δεν ξέρει το Αφγανιστάν. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση, πολύ περίπλοκη. Πώς μπορούμε εμεί ε, να εφαρμόσουμε τους διεθνεί κανόνες ε, στο Αφγανιστάν Πώ μπορούμε να εφαρμόσουμε και να επιβάλλουμε τα δικαιώματα των γυναικών είναι πραγματικά πολύ διαφορετική κατάσταση. Σε άλλα σημεία θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών. Ε, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για την, ε, τον αλφαβητισμό και την εκπαίδευσή τους. Κορίτσια 13 χρονών πολλές φορές δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο στις αγροτικές περιοχές γιατί δεν βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα. Απέχουν 10 χιλιόμετρα, πρέπει να περπατήσουν και τα υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας. Στερούνται λοιπόν παιδείας. Άυμα είναι αμόρφωτες, πώς μπορούμε να περιμένουμε πως θα αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους και ότι θα συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. Πολλά προβλήματα υπάρχουν. ο καρζάι μπορεί να κατηγορηθεί γιατί υπάρχει μεγάλη διαφθορά, νεποτισμός, υπάρχει ατιμορρησία, πολύ αδύναμο κράτος δικαίου. Πολλές προκλήσεις έχει να αντιμετωπίσει ο καρζάι. πώς μπορούμε να σηματοδοτήσουμε την αλλαγή, πώς μπορούμε να ολοκληρώσουμε τον πρώτο γύρο. Μεγάλη πρόκληση για την Επιτροπή, το, την εκλογική. Πώς, πόσες κάλπες ήρθαν από τα διάφορα μέρη και είναι ύποπτες Πώς μπορούν να, να, να τα μετρήσουν όλα αυτά και να τα σταθμίσουν. Μεγάλη πρόκληση, τεράστια. Ακόμα και αν αποκλειστούν κάποιες κάλπες από την καταμέτρηση, ακόμα και αν εξεταστούν οι 600 ε, ενστάσεις Κανονικά κανένας δεν μπορεί να φτάσει στο 50% συν 1. Και σύμφωνα με το Σύνταγμα περνάμε σε δεύτερο γύρο. Αλλά θα πρέπει να το δεχτούμε. Αυτή είναι η αρχή της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν δεν βγάλει κανένας 51%. Κατάσταση τώρα της νομοθεσίας στο Αφγανιστάν. δεν συμφωνεί με τις διεθνείς ε, συνθήκες. Το Αφγανιστάν έχει υπογράψει έξι Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα ε, των ε, Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Μόνο αυτή η συνθήκη δεν έχει επικυρωθεί. Οι υπόλοιπε έχουν όλες επικυρωθεί. Να τονίσω πως όταν συντάχθηκε το Σύνταγμα και τέθη προσυζήτηση το 2004, στο τέλος του 2004 νομίζω, υπήρξε μεγάλη συζήτηση για να γίνει δεκτό αυτό το άρθρο διεθνώς. Η νομοθεσία του Αφγανιστάν θα πρέπει να συμφωνεί, ή να είναι σύμμορφη προς τη διεθνή νομοθεσία. Αλλά σε εκείνο το άρθρο λέει ότι καμιά νομοθεσία δεν μπορεί να γίνεται που να είναι σε αντίθεση με τις Ισλαμικές αρχές. Και τα δυο άρθρα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έρχονται διαρκώς σε αντιπαράθεση. Νέα νομοθεσία. Οικογενειακό δίκαιο. Πολύ σοβαρή νομοθεσία. Το έχω συζητήσει στο Υπουργείο και με το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έθεσε αυτό το θέμα στην ε, κοινωνία των πολιτών. Και τελευταία έκαναν κάποιες προτάσεις. Ακόμα και αυτό το θέμα Αυτός ο νόμος θα υποβληθεί, θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο. Ποια είναι η θέση σας, τους ρωτήσαμε, αλλά δυστυχώς κανένας δεν το πήρε σοβαρά. Μετά που πέρασε από το γραφείο του Υπουργού και έφτασε στο Κοινοβούλιο, τότε προέκυψαν όλα τα προβλήματα. Και το πρόβλημα είναι πως το Κοινοβούλιο είναι περισσότεροι οι συντηρητικοί βουλευτές που ακολουθούν και αγωνίζονται για το Ισλάμ. Ναι, ναι, τελειώνω, ολοκληρώνω. Η κατάσταση στο Αφγανιστάν όπως σας είπα, είναι ότι τελικά αφού έφτασε στο Κοινοβούλιο, ασκήθηκε πίεση από την κοινωνία των πολιτών, αφού είχε εγκριθεί πια ο νόμος, ώστε να τον ε, τροποποιήσει ο Πρόεδρος. Έχουν αφαιρεθεί πολλά άρθρα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες. Εμείς από, τις Επιτροπέ, από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν συμφωνούμε με αυτόν τον νόμο. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για πολύ παραδοσιακή και συντηρητική μουσουλμανική κοινωνία. λένε ότι υπάρχει αυτό στο Άγιο Κοράνι. Δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε αυτό από το Άγιο Κοράνι. Πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία είναι αντίθετα με τη διεθνή νομοθεσία και πολύ σημαντικά στοιχεία έχουν ήδη αφαιρεθούν και στην Επιτροπή μας, που είναι ο βασικός που διαρκώς επιμένει ώστε να βελτιώνεται η κατάσταση. Έχουμε στείλει ε, ε, επιστολές επί επιστολών στους συντάκτες ε, της νομοθεσίας. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει να συνδυαστούν μεταξύ τους ώστε να αποφέρουν καρπούς. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ, ε, αν μπορείτε να είσαστε, κύριε Λάγκαρη, ε, κάπως πιο σύντομος. Ε, όταν ξαναλέω το λόγο τώρα, κυρία Ρίζερ, έχουμε το θέμα των εκλογών. Εάν ο δεύτερος γύρος των εκλογών, εάν λάβει χώρα, μήπως θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς τη ζνοθεία, χωρίς τη βία, χωρίς να το παραδώσουμε, εκλογές του Ταλιμπάν. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, θα είναι δύσκολο ε, θα είναι δύσκολο, δύσκολο να τα καταφέρουμε. Τώρα, εάν οι εκλογές αντικατοπτρίζουν την αλήθεια, τη θέληση του λαού, είναι το θέμα βέβαια του 50% ή όχι. Χρειάζεται δεύτερος γύρος. Αυτή είναι η μεγάλη απορία μας και το θέμα αν η Επιτροπή Ενστάσεων μπόρεσε να αντιμετωπίσει και να χειριστεί τα θέματα της νοθείας. Όχι. Δεν έχει τους πόρους ούτε ανθρώπινους ούτε οικονομικούς για να το κάνει αυτό. Και γι' αυτό και δεν πήγαμε κάτω το 50%. Να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. τη δίκαιο πρέπει από τώρα να τα σκεφτούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει το χρόνο, το περιθώριο, η διεθνής κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν περάσουν δύο-τρεις μήνες, να αναλύσει τα αποτελέσματα. Για τους παρατηρητές, για την αποστολή μας, πάρα πολλά θέματα. Καλά, το παίρνω πίσω αυτό που είπα, ότι είπαμε, τα τα είπαμε όλα πολύ πιο ρόδινα, αλλά ήταν η πολιτική απόφαση, αλλά δεν ήταν μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ. Τα έλεγε στην αρχή, πάρα πολύ ρόδινα είναι για το, για, το, για το επίτευγμα των εκλογών. Ότι τα Λίμπανα πέτυχαν να ε, ε, διαταράξουν τι εκλογέ. Όταν είχαμε όμω 300 επιθέσει στη χώρα, ε, τότε δεν είμαστε αξιόπιστοι. Δεν θέλω να δώσω, δηλαδή στον κόσμο την ε, σκοτεινή, απεσιόδοξη εικόνα των πραγμάτων όπω έγινε. Όμω, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε και την αξιοπιστία τη κοινότητα και τη δημοκρατία στη χώρα. Όσον αυτό τώρα τα ΜΜΕ, προσπάθησε η κυβέρνηση να αφημώσει τα ΜΜΕ όσον αφορά τα ρεπορτάζ για την βία. Συνδύσαν 14 δημοσιογράφοι ε, γιατί ήταν κοντά στις βομβιστικές ε, πόπειρες. Ε, κάποιοι δημοσιογράφοι χτυπήθηκαν από αστυνομικού όταν προσπάθησαν να μεταδώσουν τις ειδήσει. Και βεβαίως Υπάρχουν καταγγελίε ότι τα κρατικά μέσα μερολήπτησαν υπέρ τη αποχωρούσα κυβέρνηση. Έγινε επομένω, είπαν, αυταρχικότερη η κυβέρνηση. Προσπάθειες και λοιπά. Μεγάλη πίεση επομένω, μεγάλος εκείνο για τους δημοσιογράφου και πάρα πολύ αμφιβολικά κατά πόσον υπάρχουν ανεξάρτητα έψιλον στη χώρα. Τι να κάνουμε για τις γυναίκες, το είπε ο κύριος ε, ε, Λάγκαρη. Όσον αφορά τη φίτηση στο γυμνάσιο, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στην πρωτοβάθμια. Γιατί στο γυμνάσιο πάνε από την πρώτη λίγη και μετά μόνο 4% ε, των κοριτσιών. Τελευταίους μήνες πάντως σημειώθηκε κάποια βελτίωση όσον αφορά τα δικαιώματα των ε, γυναικών αλλά και των ε, επιθέσεων έχουμε τώρα λιγότερες ε, τραυματισμούς. Και πρόκειται για κάποιες διρεκτίβες, κάποιες οδηγίες που εκδίδονται. Ε, παίρνει πάντως ε, κάποιο χρόνο μέχρι να υλοποιηθούν αυτές οι οδηγίες, αλλά πάντως είχαμε λιγότερα επεισόδια, λιγότερες επιθέσεις κατά προσώπων και άρα λιγότερους θανάτους. Βελτίωση. Πρόεδρος, και τώρα θα συνεχίσουμε, θα δώσουμε τώρα το λόγο για πάρα πολύ λίγο Ε, στον εκπρόσωπο του δικτύου ανάλυσης του Αφγανιστάν. Ε, έχετε λάβει την έκθεσή μας όσον αφορά το τι έγινε στις εκλογές, ε, δηλαδή την έκθεση που εμείς έχουμε συντάξει. τις ε, λαθροχειρίες, τις νοθείες και την υπόθεση του πώς θα πρέπει να το αποτέλεσμα προσπαθούμε να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των λαθροχειριών ότι πρώτα πρώτα είχαμε κάποιες χειριστικές κινήσεις κάποιες λαθροχειρίες που δεν είχαν ε, ε, επίδραση στο αποτέλεσμα αλλά είχαν επίδραση στον κόσμο όσον αφορά δηλαδή κάποιους υπαλλήλους οι οποίοι, ε, οι οποίοι προσπαθούν να παραπείσουν τους ε, ψηφοφόρους τι θα ψηφίσουν και από την άλλη μεριά έχουμε άλλες χειριστικές τέτοιες κινήσεις σε σχέση με άμεση επίδραση στο αποτέλεσμα πάνω δηλαδή στις ψήφους, πάνω στα ψηφοδέλτια, πάνω στι στις κινήσεις που γινόντουσαν, τις αθροχειρίες πάνω στην κάλπη και για την κάλπη. Ε, σήμερα συζητήσαμε και για τους διεθνείς παρατηρητές. Ε, πάρα πολύ λίγοι παρατηρητές ε, μπόρεσαν να παραστούν εκεί που είχαμε μαζικές λαθροχειρίες. Ε, ε, πάρα πολλά γίνανε το βράδυ πριν τις εκλογές ή αμέσως μόλις έκλεισαν τα εκλογικά κέντρα. Οπότε οι αρχικές ε, εκθέσεις, οι αρχικές αναφορές των παρατηρητών δεν μπόρεσαν να περιλάβουν αυτά τα περιστατικά. Ακούστηκε πριν κάτι για τις ψηφοφόρους, τις γυναίκες. Ε, Έχουμε ολόκληρη έκθεση που ασχολείται με τις πλασματικές ψηφοφόρου, ψηφοφόρου φαντάσματα. Και είναι σίγουρο ότι ο αριθμό των 17 εκατομμύρια που ελέγχθη για ψηφοφόρου είναι κάτι το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό, δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια. Πρώτα ευχαριστούμε πάρα πολύ μεστά τα σχόλιά σας και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις προσεκτικά. Τώρα έχω και άλλους ανθρώπους που το λόγο. Ο Μπιός, Νίλσεν και άλλοι. Äh, ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης πολύ για τις πολύ ειλικρινείς και ανοιχτές ε, παρατηρήσεις σας και τις επικρίσεις βέβαια εις βάρος του στρατηγού Μοριγιών κατανοητές διότι είχαμε διαβάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι δυσκολίες είχατε. Για τον κύριο Λαγκάρη λοιπόν πρώτα. Ακούσαμε πολλά για τις ανισότητες που επιβάλλει ο νόμος σφάρος ε, των γυναικών. Τι θα λέγατε λοιπόν εσείς ως, ε, το, προς το θέμα αυτό, τι μπορεί να διορθωθεί ακόμη, τι προβλήματα επισημαίνετε ως προς τις αδυναμίες της δικαιοσύνης στο Αφγανιστάν και επίσης τι νομίζετε ότι μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Ευχαριστώ. herra hyvä. Ευχαριστούμε για τώρα κύριε Σομπιόλ, το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Όμω θα ήθελα να σα πω το εξή. Στην μέση διάταξη δεν προβλέπεται να συζητήσουμε μόνο για τι εκλογέ στο Αφγανιστάν. Απλώ προβλέπεται να συζητήσουμε γενικότερα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό ακριβώ θέλω να σα πω ότι όλα όσα εσεί μα είπατε, όλα όσα μα διευκρινίσατε, όσα μα αναλύσατε, όλα όσα είπατε ήταν πάρα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και δεν δε, δε, θέλω να ξεχωρίσω καμία παρέμβαση σαν πιο καλή από τις Όλα όσα είπατε μας ε, βοήθησαν να καταλάβουμε καλύτερα το τι έγινε και το τι γίνεται σε σχέση με τις ε, εκλογές των Παρχικών Συμβουλίων αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν τις προεδρικές, τις κοινοβουλευτικές τώρα. Κάτι άλλο για αυτό το ερώτημα. Το... Όταν μιλούμε για θέματα δικαιώματα, τι εννοούμε. Δεν θα πρέπει όλα να τα σχετικοποιούμε και να θα κάποιες ε, αξιολογικές κρίσεις ε, θρησκευτικέ, πολιτιστικές ε, και έτσι να διαφοροποιούμε τις παρανθρώπινες αυτές αξίες χώρα. Όμως έχουμε κάποιες προτεραιότητες, να είναι ξεκάθαρες ποιες είναι οι προτεραιότητες για κάποια χώρα. Για κάποια χώρα που που, που, που πάσχει, που είναι ασθενής, που είναι λαβωμένοι. Και αυτό δεν είναι σχήμα ρητορικό, φυσικά. Και νοσεί το Αφγανιστάν. Ε, μέσα στην ιστορία του τώρα πάσχει ε, αυτούς όλους τους ε, πολέμους όμως υπάρχει κάτι άλλο πολύ πιο συγκεκριμένο από πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για άντρες και για γυναίκες και εκεί πάσχει αυτή η χώρα Πολύ μεγάλο τμήμα της χώρας πάσχει. Και Αγγόλα και Σιέρα Λεόνα. Μιλούμε για τις χώρες που έχουν το ρεκόρ της παιδικής νησιμότητας. Αφγανιστάν και αυτές οι δύο χώρες. 152 ανά χίλια παιδιά που γεννιούνται πεθαίνουν και έχουν τέλο πάντων κάποιε μολυσματικέ ασθένειε που έχουν πλήξει περίπου τα, τα μισά παιδιά. Υποσυντισμός χρόνικος, χρόνιος. Και μέσω ζωής, μέσα στη διάρκεια ζωής 43 ετών. Οπότε βλέπουμε που είναι το, το θέμα στη χώρα. Ο κ. Λαγκαρή είπε κάτι που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Όπως και να αξιολογούμε τα πράγματα από πολιτική πλευράς, έχουμε την διεθνή παρουσία που παρατείνει την παραμονή της στο Αφγανιστάν. Πρέπει ότι αυτό είναι θετικό, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Και άρα θα πρέπει να θέσει κάποιες προτεραιότητες αυτή η διεθνής ε, παρουσία στο Αφγανιστάν. Ο διεθνής παράγων εκεί με τι θα ασχοληθεί. Όχι βέβαια. Μόνο καταπολεμώντα του Ταλιμπάν που τους εξομοιώνουμε του τους ε, τρομοκράτες. Όχι, χρειάζεται ε, μια άλλη αντιμετώπιση. Χρειάζεται αγώνες για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. ορισμένο, δηλαδή προς το ιατρικό, προ το, προς, το, προς το πώς θα δώσουν προτεραιότητα ας πούμε όχι στις σφαίρες αλλά στα εμβόλια. Αυτό ήθελα να τονίσω. Η κατακλείδη νομίζω ότι αυτό θέλει και ο κόσμος στο Αφγανιστάν. Η Διεθνής Επιτροπή του Βαριστρού Σταυρό έκανε κάποια έρευνα για τα δικαιώματα και οι περισσότεροι Αφγανοί είπαν ότι θέλουν πρώτον φαΐ, δεύτερον προστασία κατά της βίας και τρίτον θέλουν να μπορούν να έχουν κάποιο είδους ε, ιατρική κάλυψη. Πες τον Αύγουστο είχαμε την διάσκεψη στο Παρίσι, διάσκεψη των δωρητών. Και εκεί πέρα καταρτίστηκε ένας πίνακας των ε, προτεραιοτήτων όμως, πουθενά δεν αναφέρθηκαν τα ιατρο-υγειονομικά θέματα. Αυτά αναφέρονται έτσι, θεωρητικά μόνο. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει το ε, τουρκικό νοσοκομείο, το τελικό νοσοκομείο, το νοσοκομείο Ιντιραγκάντι. Δηλαδή γίνεται κάποια προσπάθεια προς αυτή την ε, κίνηση. Και επίσης υπάρχει μια τάση εξαφγανισμού. Προσοχή, θα πρέπει για τα ανθρώπινα δικαιώματα πάλι να δώσουμε τέτοια κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Κλείνουμε τώρα τη συζήτηση και θα, ε, μάλλον ε, έχουμε ακόμα ένα σημείο πολύ σημαντικό στην ημερήσια διάταξη και θα ήθελα να έχουμε λίγο χρόνο για να το εξετάσουμε. Ναι, εντάξει, θα μιλήσω για γίνεται πιο γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. τα αμερικανικά στρατεύματα και τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ θα πρέπει να περιορίστουν στο να προστατέψουν τον αυγανικό πληθυσμό. Εμεί έχουμε παρατηρήσει, έχουμε γίνει μάρτυρες σε πολλά ε, θύματα όπλων. Ο πρόεδρος Σαρκοζή, η Άγγελα Μέρκελ, ο Γκόρντον Μπράουν θέλουν να διοργανώσουν μια διάσκεψη για το Αφγανιστάν ώστε να αναπτύξουν μια προοπτική για να μπορέσουν να δώσουν στον αφγανικό λαό την ευθύνη. Με αυτό με αυτή τη βάση θα ήθελα να σας ε, θέσω το εξής ερώτημα, αφού σας ευχαριστήσω για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι... σε ποιο βαθμό μπορούμε να περιμένουμε αυτές οι δηλώσεις να έχουν ε, αντίκτυπο στο Αφγανιστάν. Μπορεί να έχουμε ένα δεύτερο γύρο, μπορεί και όχι. Ποια είναι η προοπτική. Μπορούμε να μιλήσουμε για ελεύθερες εκλογές στο νότιο Αφγανιστάν. Διότι στο Αφγανιστάν πολιτικές αρχές περιορίζονται γεωγραφικά στο κέντρο και στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ποια είναι η δική σας άποψη, την άποψη δηλαδή των ε, οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να επανέλθω σε ένα ερώτημα στο οποίο ίσως να είναι δύσκολο να απαντήσετε κυρία Αγκαρή. Εσείς αναφέρατε πολύ, μάλλον και αναφέρθηκε πολύ, η βία που ασκείται και που φόβησε τους εκλογείς και τους εμπόδισε από το να μεταβούν στα εκλογικά κέντρα. Αλλά ήθελα επίσης να σας ε, μιλήσω για την απογοήτευση των Αφγανών όσον αφορά τα θέματα πρόσβαση στην παιδεία, στην υγεία, στην κατάρτιση, στην απασχόληση. Εγώ είχα τακτικά την ευκαιρία να ανταλλάσσω απόψεις με νέους Αφγανού στη Γαλλία. Αυτούς τους νέους που επέλεξαν την μετανάστευση για να προσπαθήσουν να επιβιώσουν. Ακριβώς μας είπαν αυτά τα πράγματα. Μας λένε φεύγουμε από το Αφγανιστάν γιατί δεν μπορέσαμε να έχουμε πρόσβαση στην παιδεία, δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει δουλειά, τίποτα. Και λίγο μιλάνε για τους ε, Ταλιμπάν και για τη βία. Έχω δύο-τρία πράγματα να σας πω. Θα πάω πολύ γρήγορα. Επίσης, δεν φοβάστε μήπως η σύσταση της επόμενης κυβέρνησης, αν δυστυχώς και το φοβηθώ, φοβάμαι, υπάρχουν ακόμα πρώην ε, κλιματίες πολέμου, διάφοροι διεφθαρμένοι αυλικοί και εμπόροι ναρκωτικών σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν φοβάστε ότι το γεγονός ότι αυτές οι εκλογές γίνονται υπό την κάλυψη της νομιμότητας μιας εκλογικής διαδικασίας που έγινε υποτίθεται ε, υπό την διεθνή εποπτεία αποθαρρύνει τελείω τον πληθυσμό. Και όταν ο πληθυσμό αποτελείται από 60 μέχρι 70% από νέου, ποιο είναι το όραμα για το μέλλον που προτείνεται σε αυτόν τον πληθυσμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας δώσω το λόγο για δύο λεπτά κύριε Λαγκάρε και μετά θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσης διάταξής μας. έχετε το λόγο. Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η ίση πρόσβαση από τους ε, υποψηφίους στις εκλογές. Όλοι αντιπροσωπεύθηκαν σωστά, εκπροσωπήθηκαν σωστά, δόθηκε ο ίσος χρόνος σε όλους τους υποψηφίους, η τηλεόραση διευκόλυνε τις συζητήσεις, ακούστηκαν διάφορες απόψεις ε, και ούτω καθεξή. και βέβαια για τη διαφήμισή τους έπρεπε να πληρώσουν το κόστος. Τα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης κατηγορήθηκαν ότι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο προς όφελος ενός μόνο υποψηφίου. Εάν η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το πλάνο ειρήνης και συμφιλίωσης, εμείς δεν αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα της ε, ε, συμπερίληψης των εμπόρων ναρκωτικών στην μελλοντική κυβέρνηση ή των πολεμάρχων. Μεγάλη πίεση έχει ασκηθεί στην κυβέρνηση του Αφγανιστάν ώστε να εφαρμόσει το εθνικό πρόγραμμα δράσης και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κάνει πολλά και τώρα θα ολοκληρώσει την ε, προσπάθεια καταγραφής ε, των συγκρούσεων Είναι επίση προφανέ ότι οι διεθνεί δυνάμει θα πρέπει να υποστηρίξουν ε, την ανάληψη των ευθυνών από πλευρά του Αφγανιστάν και των ε, αρμόδιων του οργανισμού. Τελείωσαν τα δύο λεπτά. Παρακαλώ, συντομεύσατε. Διακόπτη, πρόεδρο. Θα πρέπει όντω όλα αυτά να γίνουν. Επίση, η δυνατότητα εκπαίδευση των γυναικών είναι πρόβλημα τα αθώα θύματα, άοπλα θύματα αναφέρθηκαν εμείς και όλες οι οργανώσεις που βρίσκονται επιτόπου τόπου, πιέζουμε τις διεθνείς ε, δυνάμεις που βρίσκονται επιτόπου τόπου, ώστε να περιοριστούν τα θύματα Το θέμα της μετανάστασης, ναι, αυτό έχει συμβεί όντως. Διότι δεν υπάρχει κατάλληλη δυνατότητα για τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν στα πανεπιστήμια. Υπάρχει και πρόβλημα οικονομικό. Και η ασφάλεια επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Οπότε τα παιδιά θέλουν να φύγουν. Ε, Μελλοντική κυβέρνηση. Ναι, όντω επιδεινώνεται λοιπόν η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια. Πολλές φορές ε, βλέπουμε και ε, προβλήματα λόγω των διαφόρων ε, οπλαρχηγών και μπόρων αργοτικών. Στη νότια περιοχή του Αφγανιστάν αυτή ελέγχεται από τους Ταλιμπάν. Το 1 τρίτο της χώρας είναι υπό τους Ταλιμπάν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να διακόψουμε τώρα γιατί έχουμε μόνο μισή ώρα για ένα ακόμα πολύ σημαντικό θέμα, μια πολύ σημαντική μελέτη για τα βασανιστήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Ρίντ, εξ ονόματος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας εύχομαι ε, κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και πραγματικά επιθυμώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Κομισιόν να λάβουν υπόψη τις σημαντικές πληροφορίες που μας ε, δώσατε και θα ήθελα να σας δω σύντομα ξανά στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εν τέλει να αναφέρω ότι ο στρατηγός Μοριών, ο επικεφαλής της ε, αποστολής των παρατηρητών στο Αφγανιστάν, εκλήθη στο Κοινοβούλιο, αλλά μας ενημέρωσε ότι δεδομένης της ε, κατάστασης, όπως έχει τώρα, δεν μπορεί να απελευθερωθεί για να έρθει μέχρι ότου ε, διευθετηθεί η κατάσταση. Η Επιτροπή των Εξωτερικών, η Επιτροπή Ανάπτυξης θα εξακολουθούν να συναντιούνται φυσικά μαζί του, όπως και με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν. Θα έχουν την ευκαιρία συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου να τον συναντήσουν. Ευχαριστώ και ας τώρα, ας παραδώσω μάλλον τώρα το λόγο στον πρώτο αντιπρόεδρο, κύριο Ζήπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως προβλέπει το πρόγραμμά μας, στο σημείο 5 τώρα έχουμε να συζητήσουμε μία μελέτη σχετική με τα βασανιστήρια Εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Μακάρθη, Αναλένα Σβένσον Μακάρθη, για την παρουσία της εδώ και μπορώ να δώσω το λόγο. Μακάρι να μπορούσα να σας δώσω για πιο πολύ από 10 λεπτά, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε περιθώριο. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να περιοριστείτε κι εσείς με βάση το χρονοδιάγραμμα. Από ό,τι μάλιστα έμαθα ο κύριος Πισάρα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Θα τον παρακαλέσω λοιπόν να λάβει το λόγο ύστερα από εσά. Κυρία Σασόν Μακάρθη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα προσπαθήσω να είμαστε δυνατόν πιο σύντομοι. Ευχαριστώ καταρχά που με καλέσατε σε μια ανταλλαγή απόψεων για το έγγραφο εργασία, ενημέρωση καλύτερα και θα ήθελα επίση να ε, συγχαρώ και τα μέλη εδώ της Επιτροπής για την εκλογή ή επανεκλογή τους. Ο στόχο αυτού του εγγράφου ενημέρωση που σα παρουσιάζεται σήμερα είναι η παρακολούθηση τη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των βασανιστήριων και τη ε, της κακομεταχείρισης από την δημοσίευση μια ευρύτερη μελέτη που είχαν αναθέσει οι προκάτοχοί σα και που αναλάβαμε μαζί με την OMCT, καταθέσαμε τον Απρίλιο 2007 και παρουσιάσαμε τον Δεκέμβριο πέρσι στην Επιτροπή σα. Αυτή η μελέτη έχει διάφορες, ε, περιείχε μάλλον διάφορες συστάσεις και παρατηρήσεις για ελλείψεις και οπισθοδρομήσεις ή προβλήματα που ε, σημειώνονταν. Λοιπόν, μια και δεν έχουμε χρόνο, ε, δεν είχαμε χρόνο, αποφασίστηκε να μην γίνουν ε, επισκέψεις επιτόπου και έτσι ε, μόνο με βάση το ερωτηματολόγιο που αποστήλαμε στα κράτη-μέλη συστάθηκε η δεύτερη αυτή έκθεση σχετική με την Αλγερία, την Μπαγκλαντές, τη Γεωργία, την Αιγύπτο, το Μαρόκο, την Ουκάντα και την Ουκρανία και αποφασίστηκε επίσης η αποσταλή ερωτηματολογίου και σε σε αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπροσωπείες όπως η παραδείγματι ε, σχετική με τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι με βοήθησαν και στην επίσκεψή μου στους Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο φέτος και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την ενημέρωση που μου διέθεσαν πολύ γρήγορα πολλές φορές χωρίς δηλαδή επαρκή χρόνο προετοιμασίας. Χωρίς τη βοήθειά του, θα μπορούσα να έχω συντάξει το κείμενο αυτό. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θα μιλήσω πρώτα, μετά για το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χωρίς τα κράτη-μέλη. Ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναμφίβολα προσφέρει πολύτιμη καθοδήγηση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαι πεπισμένη ότι κατά τη διάρκεια της νέας αυτής θητείας ε, η ισχυρή φωνή του ε, Κοινοβουλίου και της Υποεπιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα συνεχίσει να αντιχεί και να συμβάλλει ε, για να εξασφαλιστεί ε, συνεπής αποτελεσματική και ουσιαστική βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γέννη με βάση την ευρωπαϊκή πολιτική. Σημαντικό λοιπόν συμπέρασμα από, το, από τη μελέτη μου, συγκρινόμενα η κατάσταση με την προηγούμενη περίοδο, δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση, γνώση, καλύτερη γνώση των κατευθυντήριων γραμμών σχέση με, τα, ε, με την κακομεταχείριση και τα βασανιστήρια και άρα έχει δράσει ως καταλήτη στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν προκειμένου τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και Κατ' Ορμελών. Συνίσταται λοιπόν να συνεχίσει αυτόν τον καταλητικό ρόλο το Κοινοβούλιο και να αναλάβει και την ε, συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθυντικών γραμμών προς το τέλος του 2010-2011 με βάση τις γραμμές που προσδιορίστηκαν ήδη και επίσης προτείνεται να ε, διατυπώνουν διαρκώς ζητήματα σχετικά με, τις, με τα βασανιστήρια και τις, ε, την κακομεταχείριση οι ευρωβουλευτές στις παρατηρήσεις τους, στις συναντήσεις τους, επαφές ή αποστολές σε τρίτες χώρες ιδιαίτερα και ενδιαφερομενα κάτι κράτη-μέλη ή εμπλεκόμενα κράτη-μέλη. Για το Συμβούλιο, πρώτη θετική πτυχή ασφαλώς είναι η αναγνώριση της αναθεώρησης της ενημέρωσης των κτηριών γραμμών. Ιδιαίτερη ε, σημασία και ενδιαφέροντο στα νέα μέτρα, στην εφαρμογή των μέτρων, ήταν η σύσταση ε, προ τι ε, τρίτε χώρε για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών δράσεων, αναχώρα δηλαδή, με τις 12 προτάσεις, σύμφωνα με τι 12 προτάσει που είχαμε υποβάλει και το Δεκέμβριο του 2007. Επίσης υπάρχει υποχρεωτική ε, κατάρτιση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα τώρα για οποιονδήποτε συμμετέχει σε αποστολές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο εξωτερικό, για τους υπαλλήλους δηλαδή. Και επίσης ενσωματώνεται η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες όλες της Ένωσης, πράγμα το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί ασφαλώς και στο μέλλον. Αυτά λοιπόν είναι τα θετικά. Από την άλλη, σημαντικό πρόβλημα το οποίο επεσήμαναν αρκετοί παράγοντε με του οποίου μίλησαμε στις Βρυξέλλε, ήταν η έλλειψη συνέπεια και αποτελεσματικότητα ω προ την πολιτική για την αποτροπή των βασανιστήριων και τη κακομεταχείριση. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι αφού είναι τόσο περίπλοκη η κατάσταση και τόσο περίπλοκη η καταπολέμηση των βασανιστήριων και τη κακομεταχείριση, θα πρέπει το Συμβούλιο να δείξει περισσότερη συνέπεια. Έτσι, συνίσταται η άτυπη τώρα task force για τα βασανιστήρια να αναβαθμιστεί σε επίσημη ομάδα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζουμε το 2008 είχε την εκστρατεία, είδε την εκστρατεία της Εθνούς ημέρας για την υποστήριξη των θυμάτων της, ε, των βασανιστήριων. Εξαίρετη πρωτοβουλία η οποία βοήθησε ιδιαίτερα τις ε, διάφορες αντιπροσωπείες, 70 αναπατώμε, να αναπτύξουν δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και στα τρίτα κράτη. Εξασφάλισε κονδύλια και από διάφορους οργανισμούς και σώματα για εκδηλώσεις, όπως παραδείγματι την 60 την ερωτασμό της 60ης επαιτίου της Οικουμενικής Διακήρυξης των Σπουδών Δικαιωμάτων. Αλλά συμπληρώνω ότι αφού δεν έχουμε επαρκείς απαντήσεις ε, στα ερωτηματικά μας, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν υπάρχει επαρκή συνεργασία ε, μεταξύ των φορέων αυτών της Επιτροπής και της Κοινωνίας των Πολιτών. Εγώ ξέρω προσωπικώς ότι υπάρχουν αρκετές καλές οργανώσεις της ε, Κοινωνίας των Πολιτών, δραστήριες και αποτελεσματικές. Προτείνουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση. Και προκειμένου θα ήθελα να φωτώ σε ακόμη δύο θέματα. Καταρχάς ότι θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να καταγράφει θετικές εμπειρίες και να τις διαθέτει στις αντιπροσωπείες ε, με μια απλή βάση δεδομένων online, βάση για τα βέλτιστα παραδείγματα. Έτσι αυτά μπορούν να αποτελέσουν και αντικείμενο συζήτηση στις επαφές των αντιπροσωπιών. Και επίσης θα προτείναμε να ενσωματώσει την ε, διάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστήριων και της κακομεταχείρισης και να προβλέψει και την υποχρεωτική κατάρτιση των υπαλλήλων της ε, όπως ακριβώς προβλέπεται και στο Συμβούλιο ενώ μέχρι τώρα είναι μόνο προαιρετική αυτή. Ας περάσω τώρα στα κράτη-μέλη. Σε διμερές επίπεδο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτα κράτη. Προτείνεται να προσδοριστούν συγκεκριμένες ε, στρατηγικές δράσεις αναχώρα και να εφαρμόζονται όποτε είναι δυνατό αυτό πολιτικά και βέβαια δίνονται κατάλληλες κατευθύνσεις και από τις παρατηρήσεις των Ηνωμένων Εθνών και επίσης υπάρχουν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές όπως η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Σπουδών Δικαιωμάτων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστήριων κτλ. Ε, πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα burden sharing, δηλαδή ανάληψης του βάρους του κόστους της ανάπτυξης τέτοιων νέων μεθόδων μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων κρατών, γιατί είναι πολύ δύσκολο για ορισμένες μικρότερες χώρες να συμμετάσχουν σε τέτοια προγράμματα, δεδομένου ότι δεν έχουν επαρκείς πόρους, ανθρώπινους ή υλικούς. Πιστεύουμε επίση ότι θα πρέπει να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη στην πιο αποτελεσματική εφαρμογή τη σύμβαση κατά των βασανιστήριων και άλλων ε, ε απάνθρωπων ε, ή σκληρών ε, μεταχειρήσεων και να αναπτύξουν μεταρρυθμιστικά προγράμματα σε τομείς, σε τομείς όπως η αστυνομία, οι δυνάμεις ασφαλείας, οι φυλακές, η δικαιοσύνη κτλ. Επίσης, σε πολυμερές επίπεδο συνίσταται να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συνεργασία της με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη και επίσης ε, σημειώνουμε ότι είναι απαραίτητο να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα κατάλληλα όργανα να παραμείνουν ή αν δεν είναι να γίνουν ανεξάρτητα γιατί υπάρχουν πολλές πιέσεις αυτή τη στιγμή. Και επίσης ε, η ε, συστάσεις των οργάνων αυτών, των οργάνων δηλαδή της συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Για να κλείσω τώρα θα ήθελα ιδιαίτερα να σημειώσω τα λόγια ενός διπλωμάτη Βρυξέλλες, ε, ο οποίος είπε ε, ότι θα πρέπει ό,τι παραγγέλνουμε στους άλλους να το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι δηλαδή ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2006 που ξεκινήσαμε να μελετάμε την έκθεση, διαρκής ε, ανησυχία που εξέφραζαν οι ευρωπαϊκοί παράγοντες, οι διεθνείς ε, οργανισμοί, η κοινωνία των πολιτών, οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, ήταν διαρκώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πληρούν τις προδιαγραφές που θέλουν να επιβάλλουν ως προς τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση σε τρίτες χώρες. Και βεβαίως είναι προφανές ότι πρέπει τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα στις δραστηριότητες της αντιμοτρομοκρατική δράσης της CIA και της ε, πτήσεις μεταφοράς κρατουμένων λαθρέα μέσω ευρωπαϊκών κρατών κάθε ε, δυνατότητα για διερεύνηση, ανάκριση, δίωξη των παράνομων δραστηριοτήτων. Δεν υπάρχει χώρος για την παραμικρή δραστηριότητα βασανιστήριων ή κακομεταχείριση στην Ευρώπη και αυτό πρέπει να το κάνουμε και για να ε, εξασφαλιστεί η βεβαιότητα ότι και οι αξιωματούχοι των ευρωπαϊκών οργάνων έχουν μέτωπο καθαρό ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως προς την ε, αποφυγή των βασανιστήριων και πάνω απ' όλα ακόμη και στις περιπτώσεις της ε, ε, καταπολέμησης Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να λέει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή την ευκαιρία που μα δίνετε για να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων τη βάση αυτή τη μελέτη. Και θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω ότι η προηγούμενη μελέτη του 2007 είχε συμβάλει σημαντικά στην διαδικασία την οποία ε, έκανε το Συμβούλιο για να αναθεωρήσει τις ε, κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βασανιστήρια. Αυτή η μελέτη κάνει πολλές παρατηρήσεις και συστάσεις που δίνουν πολύ χρήσιμες οδηγίες και πρακτικές ιδέες ώστε οι κατευθυντήριες μας γραμμές να γίνουν πιο λειτουργικές και νομίζω πως από κοινού με την Προεδρία και τα κρατημέλη προσεκτικά θα εξετάσουμε κάθε μια από αυτές τις συστάσεις για να δούμε πώς μπορούμε περαιτέρω να βελτιώσουμε τις δράσεις μας. Θα ήθελα επίσης με την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω τη σημασία που αποδίδουμε στην καταπολέμηση των βασανιστήριων ή κακομεταχείρισης, οποιασδήποτε κακομεταχείρισης, παραμένει προτεραιότητα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως είπαμε, Είμαστε ικανοποιημένοι από την παρατήρηση που λέει ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αυξημένο ενδιαφέρον και συνειδητοποίηση όσον αφορά τις κατευθύνσεις γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα βασανιστήρια στις διάφορες αποστολές και στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Αυτό είναι θετικό και έχουμε προσπαθήσει ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών κατά τη βάση των συστάσεων του Κοινοβουλίου ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση, να κάνουμε κατάρτιση, να διαδώσουμε όσο γινόταν τις κατευθυντήριες γραμμές και φυσικά δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε απόλυτα για το γενικό συμπέρασμα της μελέτης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει μια συνεπή ε, αποφασιστική καθορισμένη και αποτελεσματική δράση, ε, μια φράση που τα λέει όλα, αλλά στην καρδιά μια τέτοια φράση ε, βρίσκεται η πολιτική βούληση όλων των αρμοδίων φορέων ε, στι Βρυξέλλε, στι τρίτε χώρε, αλλά και σε όλου του ενδιαφερόμενου φορεί. Και δεν μιλά μόνο για την Κομισιένα, αλλά και για του ΜΚΟ και όλου του φορεί που μπορεί να συμβάλλουν για την πρόληψη των βασανιστήριων. Και πιστεύω πως ε, εδώ μπορούμε να δούμε ότι πρόκειται για μια συνεχιζόμενη διαδικασία και το θέμα της πολιτικής βούλησης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί όσον αφορά θέματα συνέπειας ε, και συνοχής που σωστά τονίστηκαν ως ε, θέμα κλειδί όσο και για να ολοκληρώσουμε να πω ότι καλωσορίζουμε αυτή τη μελέτη που είναι πολύτιμη συμβολή στις δικές μας προσπάθειες στην βελτίωση δηλαδή των δράσεών μας για την καταπολέμηση των βασανιστήριων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και μπορείτε να πάρετε το λόγο για συζήτηση. Ο Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη σας. Δεν με τράβηξαν ιδίως αυτές οι συστάσεις ε, για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πιο συγκεκριμένα οι συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. άμα δεν φύλαξε να το ξαναδιαβάσω πιο προσεκτικά, λέει το περί το κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο συστηματική προσέγγιση για τα θέματα που αφορούν τα βασανιστήρια, την κακομεταχείριση. Και αυτό να ισχύσει για επιτροπές και υποεπιτροπές του Κοινοβουλίου. Και σας το επενθυμίζω, η Επιτροπή μας, η Υποεπιτροπή μας, αλλά και η Διάσκεψη των Προέδρων των ε, Αντιπροσωπιών του Κοινοβουλίου είχε συντάξει στην προηγούμενη θητεία προτάσει της ε, Ελέν Φλότρο, της ε, Προέδρου τότε, ε, κάποιο είδους χάρτη πορείας, κάποιο είδους οδηγού για τις αποστολές, της αντιπροσωπείας σε τρίτες χώρες που θα αφορούσε τους συναδέλφους, τους βουλευτές. Και αυτός ο χάρτης πορείας ελάμβανε πάρα πολύ υπόψη το τι γίνεται όσον αφορά σε αυτές τις χώρες για τα προβλήματα και τα χείριση. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή διότι πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος ε, στα κείμενά μας να γυρνάμε γύρω από το ίδιο θέμα, να επαναλαμβάνουμε αένα τα ίδια πράγματα. Οπότε, προτείνω στην Πρόεδρο να αναζητήσει, να βρει αυτό το κείμενο που και επίσης είχε χρησιμεύσει και το είχε εγκρίνει και η, και των αντιπροσωπιών και αυτό το κείμενο να θεωρηθεί πάρα πολύ βασικό στοιχείο για τις ε, επισκέψεις μας. Είναι κάτι το χρήσιμο. Και κατά κάποιο τρόπο να προσέξουμε να μην το χρησιμοποιούμε ε, να μην, μην, έχουμε, μην επικαλούμεθα κάποια άλθη όσον αφορά κάποιες τέτοιες κυβερνήσεις. Όχι, θα λέμε. Συμπαθάτε με πέραν των όσων άλλων κουβεντιάζουμε, θα πρέπει δυστυχώ κάτι δυσάρεστο να σα αναφέρω. Γιατί εδώ πέρα το κοινοβούλιο μου λέει ότι υποχρεώνομαι να κάνω το και το. Γι' αυτό και σα λέω ότι αυτό το κείμενο θα ήταν πραγματικά χρήσιμο. Τώρα. Θα πρέπει να γίνει επομένω μια καινούργια γενική αξιολόγηση όσον αφορά αυτέ τι ε, βασικέ κατευθυντήριε ε, 2010-2011 πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο και γι' αυτό και θα πρέπει και η πρόεδρός μας να ε, λάβει υπόψη και αυτό το στοιχείο. Εδώ αναδύονται τα εξή θέματα. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και πολύ ε, σημαντικό και το άλλο θέμα είναι κάπως πιο γενικό αλλά και αυτό σημαντικό το πόσο αποτελεσματικές είναι οι ιστοσελίδες του Κοινοβουλίου. Εκεί όπου υπάρχει ρητή μνήμα, εκεί που ε, αναφέρονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά τα βασανιστήρια. Νομίζω ότι εκεί πέρα θα πρέπει πιο συγκεκριμένα να ασχοληθούμε και θα πρέπει και η πρόεδρός μας να ασχοληθεί ακριβώς με το πώς δεν θα ξεχνιούνται τέτοια αξιολογικά αλλά θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Επίση, σας επισημαίνω τι τελευταίε ε, γραμμές, του τελευταίου αυτού του εγγράφου που μπορεί να γίνει εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό για τον αγώνα μας. Δεν είναι δυνατόν να πρεσβεύουμε την προσέγγιση των δικαιωμάτων εάν δεν είμαστε ε, πάρα πολύ ευστηροί όσον αφορά τις ε, περιπτώσεις βασανιστηρίων τις εξαφτιστικές ε, συμπεριφορέ και πρώτα πρώτα ξεκινάμε από τα του οίκου μας μέσα στα ίσια τη Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Όχι. Αν η κυρία Σβένσον Μακάρθη έχει τίποτα να συμπληρώσει. Όχι ιδιαίτερα, Πρόεδρε. Απλώς στο πρώτο σημείο που θα θέλω να υπογραμμίσω είναι η πολιτική βούληση. Πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να κάνουμε πολλές προσπάθειες για να βελτιωθεί η κατάσταση σε μια χώρα. Χωρίς πολιτική βούληση όμως ούτε η κατάρτιση ούτε οι προσπάθειες φέρνουν καρπούς. Σε ένα από τα παραδείγματα που μελετήσαμε την Αίγυπτο επειδή η κυβέρνηση βέβαια αρέσκεται πολύ στην κατάρτιση, έγιναν, ε, δόθηκαν πολλά κονδύλια για προσπάθειες κατάρτισης ε, και από την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και από άλλες πηγές. Όμως οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις επιτόπου μας είπαν δεν κάνουν τίποτα τα χρήματα. Πρέπει να σταματήσει μάλιστα αυτή η ροή διότι δεν φέρνει το κατάλληλο αποτέλεσμα. Πολύ σωστά λοιπόν η παρατήρηση του κ. Βιόλου. Επίσης, ο οδηγός που εγχειρίζεται στους ευρωβουλευτές τις αποστολές τους στο εξωτερικό νομίζω ότι είναι πολύ καλός γιατί δείχνει ταυτόχρονα ότι και ε, η κατάσταση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το αν τη βλέπουμε από μέσα ή απ' έξω. Οι πρεσβευτές, οι διπλωμάτες στην κάθε χώρα ξέρουν ποια είναι η κατάσταση πολύ καλά. Ε, υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτερα από την Ολλανδία ή τη Σουηδία οι οποίοι ξέρουμε ότι ότι, ότι έχουν μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένω, εκείνοι έχουν καλύτερη εικόνα τη κατάσταση στην κάθε χώρα. Τίποτε πρόσφατο δεν έχω να συμπληρώσω, να συστήσω. Το πρόβλημα είναι γενικευμένο, όπω είπα, και εγώ ίδια δυσκολεύομαι να βγάλω την άκρη τώρα μόνο λίγο καλύτερα από ό,τι στην αρχή, αλλά πάντως είναι πολύ πρόσφατη η ενασχόλησή μου με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ για όποια σχόλια ακούστηκαν. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ξαναλάβει το λόγο μήπω. Όχι. Από ό,τι βλέπω. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Το έγγραφο αυτό, τα πορίσματα της μελέτης, για την εφαρμογή των κατευθυντικών γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά δείχνουν ξεκάθαρα ότι θα πρέπει το Συμβούλιο και η Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις προτάσεις, τις συστάσεις που διατύπωσε η συγγήτρια. Ήδη υπάρχει σημαντική πρόοδος, ευπρόσδεκτη πρόοδος και βέβαια υπογραμμίζουμε ότι και οι αντιπροσωπείες, ε, οι αποστολές βουλευτών ε, στις διάφορες χώρες μέλη πρέπει να γίνονται με κατάλληλη προετοιμασία της και οι βουλευτές να πηγαίνουν κάπου να, γνωρί, είναι ενήμεροι για όποια ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκδηλώνονται σε κάποια χώρα. Ήδη το έχουμε σημειώσει αυτό και ελπίζουμε να εφαρμοστεί στην πράξη τακτικά ε, ο κανόνας αυτός. Μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν οι αποστολές οι αντιπροσωπείες μας θα διατηρήσουν φυσικά ε, επαφές με τρίτες χώρες, εκ των οποίων ορισμένες έχουν και σοβαρά προβλήματα των δικαιωμάτων. Όπως επισήμανα και στο έγγραφο, υπάρχει ζήτημα ως προς την ε, ε, βοήθεια προς τα θύματα των βασανιστήριων. Κέντρα υποστήριξης που χρειάζονται περισσότερα κονδύλια φυσικά και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και σε επίπεδο γενικότερο του Κοινοβουλίου όταν έρθει η ώρα για, την, ε, για τον προπολογισμό. Για το Συμβούλιο σημειώνουμε ασυνέπεια ως προς τη δράση του, ασυνέπεια η οποία έχει ε, αντίκτυπο και στην ανταπόκριση της χώρας στόχου. Καλό θα ήταν λοιπόν να, έχουμε μια, να θεσπίσει το Συμβούλιο μια μόνιμη ομάδα εργασίας για να παρακολουθεί την κατάσταση και εν τέλει βέλτιστες πρακτικές και η ιδέα για μια ε, ιστοσελίδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία θα καταγράφονται οι βέλτιστες πρακτικές είναι νομίζω πράγματι μια πολύ χρήσιμη καλή ιδέα και οι παρατηρήσει σας, η παρατήρηση αυτού του διπλωμάτη στις Βρυξέλλες ε, είναι πολύ εύγλωτη ότι δηλαδή ε, πρέπει να κάνουμε αυτό που παραγγέλνουμε στους άλλους, αυτό που διδάσκουμε. Ε, γιατί προφανώ, εάν εμφανίζονται προβλήματα στα ανθρώπινα δικαιώματα στι δικέ μα χώρε, η ασυνέπεια θα είναι κατάφορη. Και ο καθένα ε, θα βρίσκει δικαιολογίε στη δική μας συμπεριφορά για να συνεχίσει τα βασανιστήρια. Αυτά για να συνοψίσω τα συμπεράσματα της συζήτησής μας, της μελέτης. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστώ εσάς κυρία Σφένσον Μακάρθη για, για τη δουλειά σας. Και προχωρώ στο σημείο 6 της ημερησίας διάταξης. Την αναγγελία της ημερομηνία προσεχού συνεδριάσεως που θα λάβει χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου. 3 το απόγευμα με 6.30 το βράδυ και την 1η Οκτωβρίου, έρχεται σιγά σιγά Οκτώβρης, και πάλι στις Βρυξέλλες, 1η Οκτωβρίου, 5η το πρωί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή στη συζήτηση. Ευχαριστώ τη Γραμματεία, τους προσκεκλημένους μας, τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους της Προέδρου μας και επίσης ευχαριστώ όλοι ο Πρόεδρος, ευχα... τους διερμηνείς χωρίς τους οποίους η δουλειά μας δεν θα ήταν δυνατή. Και οι διερμηνείς ευχαριστούν.